Uh, colleagues, I think we're ready to make a start, because I think most of our shadow team are here. Να, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε περισσότερο από τους σκιώδεις, ούτως ή άλλως είναι παρόντες. Να υπενθυμίσω σε εκείνους που δεν ήταν εδώ παρόντες εχθές ότι αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί. Η σειρά θα είναι. Θα ζητήσουμε από την κυρία Ρόιτοβα να μιλήσει για τις καταθέσεις εγγύησεων, για τα προγράμματα εγγύησεων καταθέσεων. Μετά θα πάμε στους γεωργικούς ελκυστήρες του κυρίου Πανζέρη και πρωτού αρχίσουμε τα οι ε, Έχουμε ενδιαφέρουσα ημέρα μπροστά μας ακόμα, ενδιαφέρον πρωινό. Είναι στην, στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας και όπως ε, ε, μπορείτε να φανταστείτε υπάρχουν κάποιοι που έχουν ξυπνήσει νωρίς και μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο. Αυτές είναι οι μόνες ανακοινώσεις για σήμερα το πρωί. προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέχεια στο σχέδιο γνωμοδότησης για τα σχέδια εγγύσεων καταθέσεων έχουν, έχουν υποβληθεί οι προτάσεις από την κυρία Ρόιτοβα. Δεν είχαμε όμως δυστυχώς χρόνο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά εκτενώς. Κυρία Ρόιτοβα, αν μπορείτε να μας παρουσιάσετε πώς έχουν τα πράγματα και θα μπορέσουμε έτσι κατά να δούμε τα θέματα. Και όταν είχαμε συναντηθεί στη μεγάλη αίθουσα πριν από κάποιες εβδομάδες που θα είχαν δύο κύριοι από πλευρά Στάιλερ, S και D, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και εσείς θα μιλήσετε εξ του κυρίου Σμιτ δεν έχουμε κανένα από τους πρασίνους ακόμα. Η κυρία δεν είναι εδώ, το κύριο Σαλβίνη. Ο κύριο Μπέγκερ νομίζω ότι την Επιτροπή είναι παρόν εντάξει, σωστό. Καλώ ήρθατε. Και θα σα ζητήσουμε να σχολιάσετε στη συνέχεια. Με ιδιαίτερη χαρά δίνω τον λόγο στην κυρία Ρόιτοβα. Την ευχαριστώ. Έχουμε αλλάξει το πρόγραμμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το δικό τη θέμα. Η κυρία Σουζάνα Ρόιτοβα έχει τον λόγο. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Και Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υψηλής ποιότητας νομοθετική πρόταση και ιδιαίτερα ικανοποιημένη είμαι από τη συνεργασία που είχαμε με όλους τους σκιώδεις εισηγητές και την βοήθεια που δόθηκε γιατί είναι ένα πολύ περίπλοκο νομοθετικό ζήτημα αυτή η πρόταση αφορά ε, τα σχέδια εγγύσεων καταθέσεων, GDS, ε, το ακρόνιμο στα αγγλικά. Θα ήθελα να πω ότι καταθέσαμε αυτή την έκθεση στα αγγλικά ως κείμενο. Θέλουμε να δούμε σε σχέση με τη μετάφραση ποια θα ήταν στα τσεχικά. Δεν ήταν εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν προβλήματα και ασάφειες. Ε, θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους να εξετάσουν και να συγκρίνουν με το αγγλικό κείμενο που χρησιμοποιούμε τις μεταφράσεις τους, διότι το αρχικό, το σωστό κείμενο, το κείμενο βάσης είναι στα αγγλικά. Πρέπει να υπάρχουν σωστές αντιστοιχίε, διαφορετικά θα υπάρξουν παρερμηνίες αν έχουν πάρει σφάλματα. Χαίρομαι που αναβάλαμε την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Αν κατάλαβα σωστά, την πέμπτη το απόγευμα θα είναι η καταληκτική προθεσμία Μέχρι τότε ελπίζω, πιστεύω ότι θα έχουμε καταφέρει να έχουμε καταλήξει σε ένα καλό συμβιβασμό. Αυτό για το οποίο κάνουμε λόγο σήμερα είναι η αναδιατύπωση μιας οδηγίας του 1994. Είναι η δική μας αντίδραση στην χρηματοοικονομική κρίση πράγμα που δείχνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας υψηλότερος ε, εναρμονισμός των όρων και λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών. Σήμερα έχουμε 40 τέτοια συστήματα εγγύησης καταθέσεων GDS που καλύπτουν διαφορετικούς κινδύνους ε, με διαφορετικούς όρους ε, και προϋποθέσεις και μπορούμε να πούμε ότι συνολικά δεν προάγονται τα ωφέλη της ενιαίας εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών. Ούτε έχουμε το ίδιο επίπεδο προστασίας ε, καταθετών. Η υψηλότερη φιλοδοξία αυτής της οδηγίας ενώ συνδέεται και με άλλες οδηγίες μέσα στο, στη δέσμη μέτρων ε, για τα χρηματοπιστωτικά, είναι ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το σύστημα θα είναι αξιόπιστο και ότι θα μπορεί να αντέξει και να μπορέσει να λειτουργήσει και σε άλλες ε, ενδεχομένως κρίσεις, πράγμα που ελπίζουμε ότι δεν θα επισυμβεί βέβαια, αλλά παρόλα αυτά. Συνέταξα κάποιες λίγες τροπολογίες ε, σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φυσικά θέλω να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Θέλω να βελτιωθούν οι πληροφορίες που διατίθενται στον καταναλωτή και θέλω οι εσωτερικές προσφορές να είναι πιο διαφανείς. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είναι τόσο δαπανηρό αυτό το σύστημα όπως φάνηκε μετά από την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διεύρυνα επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να συμπεριληφθεί και το θέμα των πιστοποιητικών καταθέσεων και βιβλιαρίων καταθέσεων που καμιά φορά αντικαθιστούν θέματα τέτοιων λογαριασμών καταθέσεων και που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα κράτη-μέλη και να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης όσον αφορά την δημοκρατία της Τσεχίας έχουμε 6.000 ε, ε, τέτοιου είδους ε, ας το πω έτσι, κεφάλαια δράσης και αν συμβεί το παραμικρό δεν θα καλύπτονται. Θα πρέπει λοιπόν εδώ στο ύψος ε, των ε, ε, χιλίων ευρώ να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό δεν θα καθιστούσε πιο δαπανηρό το σύστημα. Και είναι σημαντικό αυτό για πολλά τοπικά τέτοια, τοπικές τέτοιες πρωτοβουλίες, να συμπεριλαμβάνονται δήμοι, κοινότητες, μικρές επιχειρήσεις και πρόσωπα φυσικού ε, πρόσωπα ε, νομικού δικαίου. Θα ήθελα επίσης ε, να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να συμπεριλαμβάνονται και καταθέσεις που βρίσκονται πάνω από προσωρινά από 100.000 ευρώ. Για παράδειγμα σε περίπτωση ε, απολύσεων ή σε περίπτωση ε, απέτησης ε, ασφαλιστικών αντισταθμίσεων. Επίσης, όσον αφορά για την περίοδο καταβολής, πολλές φορές οι καταθέτες πρέπει να περιμένουν πολλές, πολλούς μήνες. Και θα πρέπει εδώ να πούμε ότι η προθεσμία είναι, όπως προτάθηκε, 10 ημέρες. Πρώτη είναι 7 ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλές χώρες, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, θα είχαν προβλήματα με αυτό. Ε, το δανέζικο και το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υποδειγματικά. Και συμφωνώ και θα έλεγα ότι πρέπει να αυξήσουμε την περίοδο εφαρμογής για αυτό το μέτρο μέχρι περίοδο 5 ετών. Μέσα σε μια πενταετή περίοδο θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν μια επτάήμερη τέτοια προθεσμία κατά ε, ε, καταβολής των ποσών στους ε, καταθέτες, ε, πράγμα το οποίο είναι καλή, καλό μαντάτο. Επίσης πρέπει να καλύπτονται σε σχέση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν διαφορετικές έδρες και υποκαταστήματα. Και αυτή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Δημοκρατία της Τσεχίας ένας, για παράδειγμα, ιδιοκτήτης έχει αρκετές, αρκετές τις τέτοιες τράπεζες ε, στην κατοχή του και δεν το γνωρίζουν πολλές φορές ε, οι καταθέτες. Πρέπει να υπάρξει η διατύπωση ότι αν έχουν καταθέσεις οι καταναλωτές σε διαφορετικές τράπεζες, αυτές οι καταθέσεις θα πρέπει να καλύπτονται μέχρι ισορίου 100.000 ευρώ. Φυσικά δεν εννοώ διαφορετικές, ε, διαφορετικά θηγατρικά υποκαταστήματα μιας ίδιας τράπεζας, αλλά διαφορετικές τράπεζες. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι τα, το σχέδιο εγγυήσεων για τις ε, καταθέσεις για το GDS ε, θα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο του συστήματος να λειτουργεί με λιγότερο δαπανηρό τρόπο. Όταν έχουμε για παράδειγμα 5.000 ε, τέτοιου καταθέτε, θα πρέπει για αυτού του 5.000 να υπάρχει ένα σχέδιο δράση και όχι για το υποθετικό σενάριο των 100.000. Και όταν γίνεται λόγος ε, για το πενταπλάσιο, όταν γίνεται λόγος για το Ταμείο ε, Εγγυήσεων για τις ε, καταθέσεις σε περίπτωση χρεοκοπίας, αυτό θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Οι καταθέτες λοιπόν δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν υπερβολικά τραπεζικά τέλη και θεωρώ ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων την ίδια προσέγγιση θα υιοθετήσουν. Ένα άλλο θέμα είναι η καλύτερη προστασία των τραπεζών. Δηλαδή, μέτρα στον τομέα της πρόληψης. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πελάτες μιας τράπεζας να μην χρεοκοπήσει, να μην πτωχεύσει η τράπεζα αν συμβεί όμω αυτό θα γνωρίζουν ότι μέχρι 100.000 ευρώ θα καλύπτονται οι καταθέσει του ε, με το Ταμείο Εγγυήσεων. Από την άλλη πλευρά, η χρήση αυτού του κοινού ταμείου για μέτρα στον ε, έγκαιρη πρόληψη και σε σχέση με την πρόταση που υποβλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ληφθεί αυτή η διαφοροποίηση υπόψη έγκαιρα σε πρώιμη φάση. Και ένα άλλο θέμα το οποίο υποστηρίζω είναι ότι τα διαφορετικά συστήματα των κρατών μελών θα πρέπει να διασυνδέονται μεταξύ τους σε διαφοροποίηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προτείνει υποχρεωτικά αυτό το μέτρο, εγώ πιστεύω ότι εθελοντικά θα πρέπει να λειτουργήσει, δηλαδή να υπάρχει διατραπεζικός δανεισμός. Το μεγάλο ζήτημα και ερωτηματικό είναι αν αυτή, αυτός ο διατραπεζικός δανεισμός είναι υποχρεωτικός, θα μπορούσε η, μια, η κρίση να μεταφέρεται από μια περιοχή στην άλλη, από μια χώρα στην άλλη. Θα πρέπει τα επιμέρους κράτη-μέλη να αποφασίζουν αν θα επιθυμούν να είναι ε, μέλη του αμοιβαίου αυτού συστήματος διατραπεζικού ε, δανεισμού. Και θα ήθελα η διατύπωση των ποσοστών κινδύνων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη να διατηρηθεί. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σύστημα το οποίο δεν θα πετύχαινε τους στόχους, διότι υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη, ιδιομορφίες, διαφορές όσον αφορά και την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό όμως που είναι σημαντικό για τους καταναλωτές είναι οι καταθέσεις όσον αφορά στεγαστικές, ε, ε, ε, στεγαστικά ταμιευτήρια να διασφαλίζονται. Μια πρόταση που θα υιοθετούσε την διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι καλύτερες δηλαδή τα καλύτερα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα θα κατέληγαν στην χειρότερη κατηγορία όσον αφορά τον κίνδυνο και θα έπρεπε εδώ να διαφοροποιηθούμε σε σχέση με την διατύπωση. Πιστεύω ότι εισάγω απλούστερες, πιο ε, διαφανείς διατυπώσεις ε, στις προτάσεις μου όσον αφορά το, τα, κείμενα των, ε, τα ενημερωτικά κείμενα στα δελτία που θα χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Επίσης, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που θα υφίστανται ε, μέσω αυτών των τραπεζικών δηλώσεων. Επίσης η γλώσσα, το γλωσσικό καθεστώς είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Και οι τράπεζες αρκετά, πολύ συχνά υποβάλλουν τα συμβόλαια αυτά σε διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα εργασίας ενός κράτους μέλους. Θα πρέπει το γλωσσικό καθεστώς λοιπόν να δούμε ότι θα μπορούσε να, αυξήσει την ε, διακρατική, τις διακρατικές επιδόσεις ε, και να δούμε το τι συμβαίνει αν ε, δεν υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες για έναν καταθέτη, για έναν πελάτη στη γλώσσα του. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Είναι εξαιρετικά περιεκτική η έκθεσή σας και εξηγήσατε και τις αλλαγές που επιθυμείτε. Τι σκέπτονται οι σκιώδεις ηγητές, η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την εισηγήτρια κυρία Ρόιτοβα Μου νομίζω ότι έχει συντάξει μια πολύ καλή έκθεση και είναι κρίμα που υπάρχουν τα μεταφραστικά αυτά σφάλματα που είπατε προηγουμένως. Να είναι η κάλυψη ανά υποκατάστημα και όχι ανά τράπεζα. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ότι η Τράπεζα της Σκοτίας και η Halifax είναι όλα, όλες οι μέλη του ομίλου Lloyds. Και όπως είπατε σωστά, πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό. Έτσι η κάλυψη θα έπρεπε να είναι ανά τράπεζα, σε μια συγκεκριμένη τράπεζα και όχι για ολόκληρο τον όμιλο. Επίσης για υψηλότερες καταθέσεις, είπατε για περιπτώσεις απολύσεων ή διαζυγίων που κάποιος χρειάζεται να μοιραστεί ένα, ένα σπίτι και ίσως το ποσό που θα μπει για πρώτη στιγμή σε έναν λογαριασμό να είναι υψηλότερο. Είναι λοιπόν οι ειδικέ περιστάσεις και όταν επισυνέβη η κρίση αυτή πολλοί έμειναν ακάλυπτοι. Εγώ τα βλέπω αυτά και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία το περιθώριο που είπατε, οι 7 των 7 ημερών, θα είναι ευκολότερο από ό,τι για άλλες χώρες. Νομίζω πάντως ότι είναι σημείο προς διαπραγμάτευση. Και η μεταβατική αυτή περίοδος μπορεί να είναι κάτι που μπορούμε να προχωρήσουμε. Άλλες χώρες θα το βρουν πιο δύσκολο. Μίλησα με τον εισηγητή της Οικονομικής Επιτροπής. Προσπαθούν να καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό γι' αυτό. Έχω εγώ έναν αριθμό τροπολογιών που έχουν πιο πολύ στόχο να κάνουν πιο συμπυκνωμένο το κείμενο και όχι να το ε, διορθώσουν. δώστε μας τη δυνατότητα να ανεβάσουμε το ποσό από τα 100.000 ή στα 150.000 ευρώ. Σας ευχαριστώ πάντως για την εργασία σας. Είναι σημαντικό νομοθέτημα. Ξέρω ότι η αρμόδια επί της είναι η Οικονομική Επιτροπή, αλλά σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, εάν καταφέρουμε να τους καλύψουμε σωστά, θα είναι πράγματι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την προστασία των καταναλωτών και για να αποφύγουμε τα όσα είδαμε να συμβαίνουν προ τριών ετών, το 2008. Ευχαριστώ κύριε Στάιλερ. Δείχνει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουμε μέσα στο παιχνίδι αυτών των ε, ε, νομοθετημάτων. Ο κύριος Κρόιτσμαν που αντικαθιστά τον κύριο Σμιτ για την, για την προστασία των καταθέσεων πρέπει να ισχύουν ορισμένε βασικές αρχές το σύστημα πρέπει να είναι στέρεο, άρα να έχει την εμπιστοσύνη των καταθετών και να αυξάνει την οικονομική σταθερότητα. Οι κανόνες θα πρέπει να είναι απλοί, δηλαδή θα πρέπει να είναι ευνόητοι για τους καταθέτες και εύκολο να εφαρμοστούν από τις τράπεζες ή τους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τα εθνικά GDS. Θα πρέπει να είναι και εναρμονισμένοι οι κανόνες αυτοί, δηλαδή θα πρέπει να διευκολύνουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ε, τραπεζικών υπηρεσιών και ίσους όρους ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων και με κατανομή του κινδύνου. Να είναι αρκετά υψηλός, ε, υψηλά τα ποσά ώστε να καλύπτουν ε, μεσαίες και υψηλές καταθέσεις, να δίνονται κίνητρα για επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλού κινδύνου και το πιο σημαντικό για μας στην ομάδα των φιλελευθέρων είναι να μειωθεί η περίοδος πληρωμών σε πέντε εργάσιμες ημέρες, όπως πρότεινε ο κ. Σίμων, στην Οικονομική Επιτροπή. Αυτό είναι σημαντικό για τους καταναλωτές, διότι η περίοδος αυτή πληρωμής είναι σημαντική για να έχουν εμπιστοσύνη οι καταθέτες στο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να αποζημιώνονται το δυνατόν συντομότερο οι καταθέτες μετά από μια πτώχευση, μια ενδεχόμενη πτώχευση και να μειωθούν στις πέντε εργάσιμες ημέρες όπως προτείνει ο κύριος Σίμψον. Και το, μεγαλύτερο, το, το ε, ε, μέγιστο όριο του Ταμείου θα πρέπει να είναι τέτοιο που να μην οδηγεί σε έξτρα συνεισφορές. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε ισότιμους όρους, ίσως όρους ανταγωνισμού γιατί ορισμένε χώρε θα ζητούν χρηματοδότηση εκ των προτέρων, άλλε θα αρχίζουν να ζητούν ε, συνεισφορέ όταν θα έχει φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο. Επίση, θα πρέπει να ζητείτε και συμβολή των ε, ε, οργανισμών που συμμετέχουν στο σύστημα. Δεν θα, θα υποστηρίξουμε λοιπόν την τροπολογία 3 για την αιτιολογική σκέψη 24. Για να χρειάζεται η νομοθεσία αυτή για να ενισχυθεί η ενιαία αγορά. Ο κύριος Σμιτ εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονό ότι η κυρία Ρότεβα στην ε, πρότασή τη δεν τονίζει την ανάγκη εναρμόνιση. Είμαστε κατά τι τροπολογία 12 επί του άρθρου 5 που δίνουν στι χώρε μέλη υπερβολική εξουσία, διότι αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα Σουηδών καταθετών σε δανέζικε τράπεζε. Για παράδειγμα, οι χώρε μέλη να μπορούν να αποφασίζουν μόνε του εάν οι τοπικέ αρχέ θα έχουν καλύτερη ε, προστασία για καταθέσεις τους σε ορισμένες τράπεζες με άλλη ονομασία και η βασική αρχή του υπολογισμού. Είμαστε κατά της ε, τροπολογίας 13 στο άρθρο 6 που αποφασίζουν οι χώρες, αποφασίζουν οι μέλη εάν θα προσφέρουν κάλυψη σε τράπεζες με την ίδια ονομασία γιατί αυτό δίνει, ανοίγει το δρόμο σε αυθαίρετο αρμπιτράζ και είναι αντίθετο με τα διδάγματα της ε, οικονομικής κρίσης. Διότι καταθέτες τράφηκαν σε χώρες με, καλύτερες, με καλύτερη κάλυψη. Για παράδειγμα, η Danske Bank στη Σουηδία, που είχε καλύτερη προστασία από τις Σουηδικές τράπεζες για ορισμένα είδη καταθέσεων. Αυτό θα οδηγήσει σε τεράστιες τρευλώσεις την ε, αγορά. Χρειαζόμαστε και καλύτερου κανόνε για την έξοδο μεταξύ των εθνικών συστημάτων. Σα ευχαριστώ. Ο κ. Φόξ, μετά η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ. Πρώτα θα ευχαριστήσω την κυρία Ρόιτοβα για την εργασία της. Νομίζω ότι έχει ακολουθήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση και χαιρόμαστε για τις προτάσεις που ε, προτείνουν ίσως όρους ανταγωνισμού για όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το να συμπεριληφθούν ε, κάποια υψηλότερα όρια καταθέσεων προσωρινά είναι σωστό, να, οδηγηθούν δηλαδή σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη οι καταθέτες. Υποστηρίζουμε και την πρόταση Ρόιτοβα οι αγορέ καταθέσεων στι διάφορε χώρε μέλη είναι διαφορετικέ και νομίζουμε ότι οι χώρε μέλη έχουν ανάγκη να έχουν ευελιξία σε ό,τι αφορά τον, τον ορισμό των ορίων. Συμφωνούμε και με την αποδυνάμωση των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του διατραπεζικού δανεισμού. Εμεί θα προτιμούσαμε να καταργήσουμε τη διάταξη αυτή απολύτω, διότι έχει επιπτώσει στην οικονομική σταθερότητα και στην εμπιστοσύνη των καταθετών και διότι δεν επιτρέπει ίσου όρου ανταγωνισμού μεταξύ όλων των τραπεζών. Χαιρόμαστε για την πρόταση Ρόιτοβα για, την, ε, για, την, για τις επιλέξιμες καταθέσεις, αλλά οι χώρες μέλη χρειάζονται μεγαλύτερη ε, ευελιξία σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, αν αυτή η χρηματοδότηση θα είναι περισσότερο εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Σε ό,τι αφορά την περίοδο ε, καταβολή των αποζημιώσεων σε περίπτωση κατάρρευση μια τράπεζα, και αυτό φαίνεται πω ενδιαφέρει του περισσότερου εδώ σήμερα, υποστηρίζουμε την πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7 ημερών ή 5 εργάσιμων ημερών. Και δεν προτιμούμε την εναρμόνιση σε 20 μέρες προτείνει η κυρία Ρόιτοβα, αν και πρόκειται για μεταβατική περίοδο μέχρι το 2015. Φαίνεται πάντως ότι οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλιστές, εμείς, ίσως και οι πράσινοι, ίσως λοιπόν δει ότι η κυρία Ρόιτοβα, η κυρία Ρόιτοβα, ότι η πλειοψηφία στην παρούσα επιτροπή είναι μάλλον υπέρ των πέντε εργάσιμων ημερών και ότι η υφιστάμενη τροπολογία δεν πρόκειται να υποστηριχθεί μέσα στην Επιτροπή μας. Αν λοιπόν πρόκειται να υπάρξει συμβιβασμό, θα προτείνω στην κυρία Ρόιτοβα να μειώσει, να μειώσει ίσως σε 10-15 εργάσιμες ημέρες και να κάνει και συντομότερη, ίσως κατά δύο χρόνια, τη μεταβατική περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε συντομότερα σε πέντε εργασίμες ημέρες. Βλέπω ότι ορισμένοι νεύουν καταφατικά. Και σε ό,τι αφορά την κάλυψη ανά brand, ανά ονομασία τράπεζας, δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι σωστό το μέτρο. Εάν κάθε τράπεζα χρειάζεται έγκριση στο Εμένο Βασίλειο, αυτό είναι έξτρα επιβάρυνση και ορισμένες τράπεζες χρειαστεί να αποσυρθούν απολύτως και δεν νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε κάποιο όφελος υπέρ των καταναλωτών. Πάντως, εργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε ευχαρίστως με την κυρία Ρόιτοβα και αναμένουμε την πορεία των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Φόξ. Άλλος κανείς. Πριν προχωρήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως σας ενδιαφέρει να σας πω ότι η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βρετανικής Βουλής έγραψε τον κύριο Μπαρόσο για θέματα ε, συστήματος αμοιβαίων εγγυήσεων και την αρχή της επικουρικότητα. Αυτά υπάρχουν βεβαίω διαθέσιμα και ίσως οι εισηγητές και σκιώδει εισηγητές επιθυμούν να τα εξετάσουν. Νομίζω ότι θα υποστήριζε κάτι τέτοιο την θέση τη κύρια Ρόιτοβα. Είναι σημαντικό πάντως να έχουμε υπόψη μας ότι και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές άλλων κοινοβουλίων στην Ευρώπη έχουν εξετάσει το θέμα αυτό. Ε, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να πάρει το λόγο, να κάνει ένα σύντομο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να εστιάσω στα πιο σημαντικά θέματα που συζητήσατε και δεν θα κάνω μια πλήρη επισκόπηση του θέματος, μια και δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την τοπική αυτοδιοίκηση και να σας ενημερώσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και γενικά το δημόσιο τομέα από το σχήμα. Ε, σχεδόν τα όλα τα κράτη-μέλη το κάνανε αυτό στο παρελθόν, όταν ε, κατάτιζαν καταλόγους για να δείξουν ποιοι καταθέτες δεν ήταν επιλέξιμοι. Τα περισσότερα κράτη-μέλη λοιπόν τότε δεν είχαν προβλέψει καμία αποζημίωση για τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών αρχών, των Δήμων και Κοινοτήτων. Οι Δήμοι και Κοινότητες έχουν εύκολη πρόσβαση στις ε, κεφαλαιαγορές. Μια και δάνεια στο δημόσιο τομέα και στις ε, τοπικές αρχές έχουν ε, έχουν προτιμησιακή μεταχείριση με βάση την οδηγία για τις κεφαλιακές απαιτήσει. Αντίθετα από ένα φυσικό πρόσωπο ή μία μικρομεσαία επιχείρηση που θα πρέπει να καλύπτονται πλήρω με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δήμοι και κοινότητε έχουν εύκολη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Επομένως δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τις, τους δήμους και τις αρχές. Για την προσωρινή Ε, νομίζω ότι είμαστε υπέρ τη υψηλότερη κάλυψη, υψηλότερο ποσού δηλαδή καταθέσεων. Η Επιτροπή σας συμφωνεί ότι επίσης ότι οι καταθέτες θα πρέπει να αποσημειώνονται μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να μην έχουν ας πούμε εναλλακτικέ ε, πηγές χρηματοδότησης για να τα βγάλουν πέρα. Τώρα, για την κάλυψη της συγκεκριμένης τράπεζας με συγκεκριμένο όνομα. Εμείς έκανα, κάναμε έρευνες και ζητήσαμε να μας πούν τις απόψεις τους οι, οι οργανώσεις των καταναλωτών. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και αμειονεκτήματα σε σχέση με την πρόταση. Ο καταναλωτής, ας πούμε, δεν θα πρέπει να ανησυχεί για το όνομα της τράπεζας που υπάρχει, ας πούμε, στο απόκομα που του δίνει η τράπεζα. Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή, όπως είπε και ένα βουλευτή ήδη, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα αρμπιτράζ και στρέβλωση των αγορών. Γιατί θα είναι μόνο δυνατόν στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, οι τράπεζες οι οποίες έχουν διαφορετικό όνομα ε, να λειτουργούν και να μην λένε στου καταθέτε ότι ανήκουν στον ίδιο όμιλο στην πραγματικότητα. Αυτό είναι δυνατόν και σε άλλα κράτη-μέλη. Συγγνώμη, δεν είναι δυνατόν σε άλλα κράτη-μέλη. Επίσης, θα μπουν σε πειρασμό οι τράπεζε, να ανοίξουν ένα τεράστιο αριθμό υποκαταστημάτων με άλλο όνομα και η όλη κατάσταση θα γίνει αδιαφανής για του καταναλωτέ. Σε 26 κράτη-μέλη, οι καταναλωτέ γνωρίζουν σε ποια τράπεζα έχουν καταθέσει τα λεφτά τους και με ποια νομική οντότητα έχουν αυτή την ε, συμβατική σχέση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό το απλό σύστημα. Μία τράπεζα, μία προστασία για τις καταθέσεις. Μόνο και μόνο γιατί σε ένα κράτος μέλος μπορεί κανείς ε, να καταθέσει σε τράπεζες με διαφορετικό όνομα που ανήκουν στον ίδιο όμιλο όμως, που είναι το ίδιο πράγμα. Ε, μετά από επαφές που είχα, ε, με διάφορου ενδιαφερόμενους. Ε, ακόμα και στον Ηνωμένο Βασίλειο μου είπαν ότι υπάρχουν αρνητικέ συνέπειες από αυτό το σύστημα. Να πω δύο λόγια τώρα για τις συνεισφορές ε, βάση του κινδύνου. Πιστεύουμε ότι αυτή, αυτό το σύστημα είναι πολύ σημαντικό. Ε, ο καταναλωτής, ο καταθέτης άμεσα δεν αισθάνεται τίποτα. Έμεσα όμως αυξάνει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και παρεμποδίζει τις χρεοκοπίες των τραπεζών. Γιατί? Γιατί οι τράπεζες πληρώνουν περισσότερα στο σύστημα ε, και αυτές που πληρώνουν περισσότερα στο σύστημα έχουν, είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Επομένως, ε, τους δίνουμε κίνητρα για να λειτουργούν ε, με ένα επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλότερου κινδύνου. Συχνά επίσης άκουσα να αναφέρετε την ε, ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά. Νομίζω θα ήταν άδικο για την ενιαία αγορά αν οι τράπεζες πλέον αρχίσουν ένα κρατός μέλος, ψήσει το άλλο κρατός μέλος Κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση. Να κλείσω με μία παρατήρηση για την πρόληψη. Δεν θα πρέπει να προάγουμε περισσότερο την πρόληψη. Η Κομισιόν έχει εντάξει στοιχεία προληπτικού χαρακτήρα. Το άρθρο 9.5 της πρότασης επιτρέπει δύο πράγματα έγκαιρη παρέμβαση. Επίσης, όλο το ποσό του συστήματος μπορούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των καταθέσεων. Άλλη προστασία. Ε, αυτό το χρησιμοποιούμε, παραδείγματος χάρη. Αν συγχωνευτούν δύο τράπεζες, ε, αν αλλάξει νομική οντότητα. Το συνολικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, μέχρι ενός ορίου. Έπειτα υπάρχει ένα δεύτερο όριο για την έγκαιρη παρέμβαση. Διαφορετικό από την περίπτωση μεταφοράς καταθέσεων. Είναι αύξηση κεφαλαίων, ε, υποστήριξη της ρευστότητας, εγγύησης κτλ. Μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι τα μέτρα που χρησιμοποίησαμε στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και οδήγησαν σε τεράστια έξοδα εις βάρος των φορολογούμενων. Η Κομισιόν πιστεύει, όπως θα ξέρετε ίσως, και θα υπάρξει μια πρόταση για τη λύση των τραπεζών, για τη διάλυση τραπεζών, ότι η έγκαιρη παρέμβαση δεν είναι κατά βιώσιμη πιστεύουμε ότι η λύση είναι το μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο θέματα. Σας ευχαριστώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ενδιαφέρουσες και χρήσιμες οι πληροφορίες. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρόιτοβα για τις τροπολογίες έχουμε ε, μέχρι τις 12 του μηνός. Στις 12 Απριλίου θα εξετάσουμε τις οπολογίες, θα, θα ψηφίσουμε στις 13. Στην οικονομικών ε, υποθέσεων θα ψηφίσουν ε, στις 9 το Μάιο. Και στην Ολομέλεια του Ιουνίου θα εξεταστεί αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ κύριε Ρόιτοβα, πολύ σύντομη στην ε, συνοψή σας γιατί δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα έπρεπε να έχει μια ισχυρή θέση ως τοποθέτηση για την περίοδο καταβολής αυτών των χρημάτων στους καταθέτες. Στη συνάντηση με τους Κιώδης πρότεινα να συμφωνήσουμε για ένα καθεστώς που θα μπορούσε να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια συντομότερη περίοδο όσο το δυνατόν πιο γοργά. Όμως ταυτόχρονα δημιουργώντας μια διαπραγματευτική θέση με την Οικονομική Νομισματική Επιτροπή με τέτοιο τρόπο ώστε να μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια θέση που δεν θα βρει αντίσταση από τα κράτη-μέλη. Και έτσι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Ίσως ε, αν είχαμε την επταήμερη προθεσμία άμεσα θα ήμουν υπέρ. Όμω αυτό θα οδηγούσε στο να μην έχουμε μια ιδανική διαπραγματευτική θέση. Γι' αυτό υπέβαλα τη δική μου πρόταση. Δηλαδή βήμα προς βήμα να συντμηθεί η περίοδος αλλά να έχουμε περιθώριο ελιγμών. Τώρα όσον αφορά Δήμου και κοινότητε, οι δήμοι οι κοινότητες δεν συνδέονται με τα θέματα των εθνικών προϋπολογισμών, τουλάχιστον σε κάποια κράτη-μέλη. Και η πρόσβασή τους στις κεφαλαϊκές αγορές δεν είναι πάντα εύκολη και γι' αυτό οι καταθέσεις τους θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον με ένα ελάχιστο ποσό, με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος στο να καταλήγουν σε μια ελληματική κατάσταση έλλειψης κεφαλαίων. Για παράδειγμα, σε σχέση με και τις, τους μισθούς των υπαλλήλων τους ε, που πρέπει να καταβάλλονται κτλ. Όσον αφορά διαφορετικά λογότυπα και διαφορετικούς τίτλους επιχειρήσεων, σε σχέση με τις δικές μου πληροφορίες, ε, οι καταναλωτές νομίζω πιστεύουν ότι σε σχέση με ένα ενιαίο νόμισμα, με ένα ενιαίο όνομα, υπάρχει διαφοροποίηση. Αν δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να υποχρεώσουμε τις τραπέζες να ενημερώνουν τους καταναλωτές πάντα για τα άλλα ονόματα και ονομασίες άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν και για το τι δεν θα καλυπτόταν. Διαφωνώ επίσης από την άλλη πλευρά με τον κύριο Σμιτ όσον αφορά την αύξηση για κατά 12 μήνες. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ε, αντέβαινε τον εναρμονισμό. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειε. Θα συζητήσουμε τι λεπτομέρειε στη συνάντηση των σκιωθών. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο Σουζάνα, για τη δουλειά που κάνατε σε αυτό το θέμα. Είναι περιεκτική και χρήσιμη η γνωμοδότησή σα. Έχουμε κάποια θέματα που πρέπει να επιληθούν. Ξέρω ότι με τη δουλειά που κάνετε και με τι τροπολογίε που θα κατατεθούν θα έχουμε ευκαιρία στι 12 Απριλίου να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Σα ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στο επόμενο σημείο και ορίζω θερμά τον κύριο Παντζέρη που είναι ο εισηγητής ε, για την, ε, το κείμενο αυτής της σημαντικής πρότασης για τους γεωργικούς ελκυστήρες. Το πρώτο που πρέπει εδώ να πούμε είναι το ότι έχουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα μετά από συζήτηση με τον εισηγητή που είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστερήσαμε την πρώτη συζήτηση και είναι μια προσωρινή έκθεση και που υποβάλλεται σε σχέση με τον κύριο Παντσέρη. Πολλά σημαντικά θέματα θα συζητηθούν υστερότερα. Από την άλλη πλευρά έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα, ένα σχέδιο για μια κρόαση. Ίσως και σε αυτό θα θέλετε να αναφερθείτε. Αυτό που θα κάνω είναι θα δώσω τον λόγο στον κύριο Παντσέρη δεν είναι τώρα η χρονική στιγμή για εκτενεί συζητήσει και για θέματα λεπτομεριών. Μετά τη συζήτηση θα έχουμε μια κρόση ούτω ή άλλω. Αν θέλει να μα δώσει την εικόνα πώ έχει το σενάριο αυτών των θεμάτων, ποιο σκιώδει είναι εδώ, η κυρία Σουλή, δεν παρίσταται. Η κυρία Ρούιλε όμω είναι εδώ. Και εγώ είμαι εδώ για του ίσια, σαν τα καταπουσιάζει. Ο κύριο Σαλβίνη όμω παρίσταται. σω λοιπόν θα θέλατε κι εσεί να συνεισφέρετε, γιατί πρέπει κάποια θέματα να τα συζητήσουμε. Ο κ. Πανσέρη λοιπόν να μας δώσει μια εισαγωγή για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και μετά θα ε, παρέμβουν οι σκιώδεις εισηγητές. Και έχουμε και τον κύριο Βόσινης νομίζω είναι, ο κύριος Βόσινης είναι από την Γενική Διεύθυνση Enterprise και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά μπορεί να μην υπάρξει χρόνος να παρέμβετε εσείς. Ο κύριος Παντσέρη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα ε, με πολύ πιο ενδελεχή τρόπο. Νομίζω παρόλα αυτά ότι είναι σαφές σε όλους ότι ο, τρόπο, ο σκοπός της πρότασης είναι να έχουμε εναρμονισμένους κανόνες για την παραγωγή των ε, γεωργικών και δασικών ε, οχημάτων, ελκυστήρων προκειμένου και ένας βασικός στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χωρίς να ξεχνάμε την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια ε, στην, της κυκλοφορίας στους δρόμους μας. Η πρόταση συνεισφέρει πέρα από την ανταγωνιστικότητα του κλάδου στην απλούστευση της νομοθεσίας για την τυποποίηση. Αυτές τις εβδομάδες είχαμε μία σειρά από επαφές με διάφορους ενδιαφερόμενους, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ομολογώ ότι προέκυψαν κάποια κρίσιμα σημεία. Δεν θα μπω τώρα στην ουσία, αλλά στις 12 Απριλίου τόσο ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία όταν γίνει συζήτηση στην ΙΜΚΟ ε, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων ε, των διαφόρων οργανώσεων να μπούμε ε, σε λεπτομέρειες. Έχουμε εντοπίσει τέσσερις κατηγορίες που θα πρέπει να τις συζητήσουμε πιο πολύ. Καταρχάς, τι θα γίνει με τη κατεξουσιοδότηση πράξης και το χρονοδιάγραμμα. Δεύτερον, υπηρεσίες μετά την πώληση. Ε, τα συνεργεία, τη συντήρηση και το θέμα της ασφάλειας. Τρίτη κατηγορία είναι τεχνικές προδιαγραφές για τις εκπομπές. Και τέλος, ε, τα οχήματα της κατηγορίας U. Για το χρονοδιάγραμμα, σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η ημερομηνία για τη θέση ισχύει είναι το 2014. Ορισμένοι έχουν αντιρρήσεις για το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές νομιθωτικές προτάσεις μέχρι το 2014 και επομένως οι ενδιαφερόμενοι ε, δεν μπορούν να κάνουν έντονες προσπάθειες ε, στα πλαίσια σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τυποποίηση. Καταλαβαίνω ότι η πρόταση τη Κομισιόν για το 2014 έγινε ακριβώ για να αποφύγουμε καταστάσει όπου θα έχουμε διαφορετικέ νομοθετικέ πράξει που παρεμβαίνουν η μία και παρεμποδίζουν την άλλη. Καλό θα ήταν να είχαμε ένα κανονισμό παρά να έχουμε πολλούς κανονισμού και επιμέρου οδηγίε επίσης παράλληλα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν συμβιβαστικέ λύσεις για να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να δημιουργήσουμε εναρμονισμένους κανόνες και τι απαιτήσει διαφο... του κλάδου ας πούμε, ε, που ενδιαφέρεται για τη διαδικασία τυποποίηση, ούτω ώστε να υπάρξει μια κάποια ανάσα σε αυτή την έντονη περίοδο μέχρι το 2014. Για το δεύτερο θέμα, τι τις ε, μετά την πώληση η πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες, κεφάλαιο 16. Αυτό ε, το κεφάλαιο 16 το αναλύσαμε και πολλοί είπαν ότι ο τομέας είναι ιδιάζοντας και η νέα πρόταση μπορεί να έχει επιπτώσεις ακριβώς στον τομέα των υπηρεσιών μετά την πώληση. Ε, και να επηρεάσει επίσης τις υπηρεσίες για τους καταναλωτές ε, σε ό,τι αφορά τα θέματα συντήρησης, συνεργείων κτλ. Θα πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία. Το θέμα της ασφάλειας υπησέρχεται εδώ που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι σε αυτόν τον κανονισμό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφάλειας. Το γεγονός ότι αφαιρέσαμε από την οδηγία για, τα, για τις μηχανές, τους γεωργικούς ελκυστήρες, δημιουργεί ένα πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας έτσι μένει εκτός του πεδίου. Εμείς ζητήσαμε από τις υπηρεσίες ε, του Κοινοβουλίου να, να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στην οδηγία για τις μηχανές και σε αυτή την πρόταση για να δούμε κατά πόσον ε, καλύπτουμε το θέμα της ασφάλειας. Τώρα, για τις ε, τεχνικές προδιαγραφές για τις εκπομπές είναι θέμα προσυζήτησης. Ένα θέμα που συζητιέται μάλιστα αφορά και το θέμα της πέδησης. Ε, συζητάμε πάρα πολύ το θέμα του ABS. Νομίζω ότι είναι πολύ αποτελεσματικό εργαλείο και για να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Ίσως υπάρχουν και άλλοι τρόποι όμως για να βελτιώσουμε την ασφάλεια που ενδεχομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και τους οποίους επομένως θα πρέπει να αναφέρουμε. Τέλος τα οχήματα της κατηγορίας U. Το θέμα αυτό ετέθη. Ετέθη το θέμα των ε, κινητών ε, οχημάτων εκτός δρόμου. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να ρυθμίσουμε. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτέ τι μηχανέ ε, εδώ. Στην πραγματικότητα αυτά δεν είναι ούτε ελκυστήρε γεωργικοί, ούτε τροποποιημένοι δασικοί ελκυστήρε. Έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Επομένω, θα πρέπει να δούμε αν θα αποκλείσουμε αυτό το τμήμα από τον κανονισμό ή αν θα πρέπει να βρούμε μία άλλη λύση, δηλαδή να προβλέψουμε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για αυτέ τι μηχανές. για, αυτά τα, για αυτή την ειδική κατηγορία γιου. Επίσης, κάποια, κάποιες ερωτήσεις που έγιναν από κάποιους ενδιαφερόμενους. Την ανάγκη ε, να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία. Ιδίως για τις ε, γουρούνες, τις λεγόμενες. Αλλά που ε, έχουν γεωργική, γεωργικό σκοπό, γεωργική λειτουργία. Και επίσης ε, άλλα μηχανήματα που τα χρησιμοποιούμε για να έλκουμε ή για να σέρνουμε. Μικρά όμως οχήματα. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια γενική σύμπτωση απόψεων ότι καλό θα ήταν να έχουμε έναν ενιαίο κανονισμό γιατί θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να πάρουμε θέση ε, στο θέμα της ασφάλειας, της οδικής ασφάλειας. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε αυτές τις εβδομάδες. Το χρονοδιάγραμμα το είπε ο Πρόεδρος, επομένως ε, αρκούν αυτά. Δεν χρειάζεται να, ε, να επαναλάβω εγώ το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Συνοψίσατε πολύ σωστά τα πιο σημαντικά θέματα. θα κάνουμε στις 12 Απριλίου, επαναλαμβάνω και εγώ, μια σημαντική ακρόαση. Ε, οι συντονιστές θα εγκρίνουν σήμερα το απόγευμα το πρόγραμμα της ακρόασης αυτής και στις 24 Μαΐ θα στείλετε την έκθεση για μετάφραση. Στις 14 έως 16 Ιουνίου θα το εξετάσουμε. Στις 6 Ιουλίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ε, θα ψηφίσουμε στην ΙΜΚΟ τον Οκτώβριο και θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ε, το χρονοδιάγραμμά σας ευθυγραμμίζεται με το χρονοδιάγραμμα εργασίας του Συμβουλίου. Σήμερα το απόγευμα έχουμε μία ακρόαση για τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες. Εκεί θα ακούσουμε διάφορα τεχνικά θέματα κτλ. Οι συντονιστές εξέτασαν, θα εξετάσουν μάλλον διάφορες προτάσεις για τεχνικά θέματα Επίσης κάποιο θέμα που ενδιαφέρει και τα μοτοποδήλατα αλλά και τις μηχανές είναι η εποπτεία της αγοράς. Να δούμε δηλαδή ποια, ποιες μηχανές δεν συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την έγκριση τύπου. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ευκαιρία στους σκιώδεις εισηγητές να προσθέσουν κάτι και ε, μου συμπεριλαμβανομένου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πλήρη συζήτηση τώρα, απλώ να δώσουμε το λόγο στου σκιώδει συζητητέ. Η κυρία Σαρτόρη που εκπροσωπεί και τον κύριο Σούλη, η κυρία Μάντια δεν είναι εδώ, ο κύριο Κρόιτσμα δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει. Εγώ, ε, εντάξει, μίλησα ω σκιώδη. Και ο κύριο Σαβίνη επίση. Κύριε Σαρτόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε το βράδυ Η ομάδα μου μου ανέθεσε να αντικαταστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Σούλη για αυτόν τον κανονισμό. Δηλαδή, μόλις τον ανακάλυψα τον κανονισμό αυτό. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Παντζέρη. Νομίζω ότι πραγματικά μας εξήγησε όλα τα θέματα που απασχολούν αυτόν τον κλάδο. Αυτά ε, εντόπισα κι εγώ σημαντικά θέματα μετά από μια πρώτη γρήγορη ανάγνωση. Καταρχάς, το θέμα της ενίας αγοράς, το ακούσαμε, όλοι συμφωνούμε. Έπειτα το θέμα της ασφάλειας και το θέμα του περιβάλλοντος. Αυτά νομίζω ότι θα είναι το νήμα που θα κατευθύνει αυτές τις ε, συζητήσεις. Επίσης το θέμα της θέσης σε ισχύ των κανόνων, αλλά αυτό το αποφασίσουμε όλοι από κοινού. Επομένω ευχαριστώ τον εισηγητή και νομίζω θα κάνουμε καλή δουλειά για το θέμα αυτό. Κύριε Κρόιτσμαν, έχετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Η κυρία Ρούλερ. Sorry. Uh, Ich ganz kurz machen. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ουσιαστικά μία πρόταση έχω. Θα έπρεπε ίσως με τον εισηγητή, τον κύριο Φάντεν να συζητήσουμε. Διότι υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις εδώ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα αυτά που θα πρέπει να εντάσσονται. Γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκυκλα για να υπάρχει καλύτερη τέτοια ρύθμιση. Δυστυχώς οι τροπολογίες, οι προθεσμίες όσο αφορά τις τροπολογίες και τα λοιπά είναι κάπως διαφορετικές, δεν εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο χρονικά. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να βρούμε όμως μια λύση για αυτό το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, οι εκπομπές ρήπων, παρότι δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο άμεσα, πρέπει να ενταχθούν και αυτές και το θέμα των πληροφοριών ανεξάρτητων συνεργείων και ε, το θέμα της ε, διάρκειας. Ευχαριστώ. Um, Mr. Ο κύριος εσείς κύριε Σαντρίνη. Όχι, εντάξει. Κάποια τελικά σχόλια από πλευρά μου υπό την ιδιότητα ω σκιώδου εισηγητού. Γι' αυτό που είπε η κυρία Ρούιλε. Αυτό το θέμα για το, τη χρονική συγκυρία είναι σημαντικό. Ανέφερε το θέμα, κύριο Σπαντζέρη, των ε, εξάτροχων και αυτό σε σχέση με τα δίκυκλα και τρίκυκλα υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ως ε, αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς ε, και χρήσεις και τελικά θα πρέπει να δούμε ότι στην κατηγορία U υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει ένας, μια απέτηση εξοπλισμού για την χρήση αυτών των οχημάτων σε οδικά δίκτυα. Αυτά θα απαιτήσουν και για το φωτισμό και για την, τον εξοπλισμό αυτών των οχημάτων κάποιες πρόσθετες απαιτήσει. Είναι απόλυτα λογικό να ζητήσουμε να υπάρξει εναρμονισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτών των θεμάτων. Κάτι υπό τη μορφή ενός παραρτήματος για παράδειγμα που θα αφορά τέτοιου είδους οχήματα. Εσείς κύριε Βασίνη σας θέλατε να τοποθετηθείτε και θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε σε λεπτομέρειες υστερότερα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αλλά ευχαρίστω να σας δώσω τον λόγο, μια και προσήλθατε. Θέλετε να κάνετε μια-δυο παρατηρήσεις, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Σε ευχαριστώ. Απλά, πολύ σύντομα, Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παντσέρη για το εύρος της πρότασης αυτής που εξετάζει με την για... όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δύο σύντομες παρατηρήσεις μόνο. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις ημερομηνίες για την εφαρμογή. Δεν έχω ειδικά σχόλια για αυτή την πρόταση. Είναι αυτή που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή βέβαια. Αλλά για την ημερομηνία εφαρμογής λάβαμε υπόψη ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να καθυστερήσουν πια άλλο. Για παράδειγμα θέματα ασφάλειας και, θα, και τα θέματα τροχοπέδησης ε, των φρένων και επίσης όσον αφορά τις απαιτήσει για θέματα όπως ε, το RMI θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τις, ε, τα μελήματα των εμπλεκομένων και των χρηστών και θα λαμβάνει υπόψη οι διομορφίες όσον αφορά τους ελκυστήρες σε σχέση με άλλα οχήματα, τις ιδιομορφίες των ελκυστήρων. Από την άλλη πλευρά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχει μια πολιτική που ακολουθούμε αυτά τα RMI να εντάσσονται μέσα στην αδειοδότηση, στην έγκριση για ε, χρήση. Από την άλλη πλευρά για το μακροπρόθεσμο πλαίσιο θα τα δούμε αυτά. Σε αυτή τη φάση αισιοδοξούμε και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και για μια νέα κατηγορία εν τέλει, ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα σε σχέση με το αν θα χρειαστούν νέες ή άλλες ε, κατηγορίες ή όχι για, την διάρκεια, για αυτή τη διάρκεια εφαρμογής. μπορώ να σας πω ότι εφόσον υπάρχουν, θα υπάρχουν απαιτήσει που θα ικανοποιούνται από κάποιες κατηγορίες οχημάτων, θα μπορούν να ενταχθούν μέσα στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού. Και έχουμε επίσης και την πρόθεση κατά τα άλλα για ότι τα δασοπονικά οχήματα ή τα οχήματα αποκλειστική χρήση γεωργία ε, να δούμε αυτέ ε, τι ανάγκε και να τι ρυθμίσουμε έτσι. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Θα δείτε φυσικά ότι η μελέτη για τις ε, Repair Maintenance Information, RME, είναι σημαντικά θέματα μέσα στο πλαίσιο του, μέσα στο οποίο πλαίσιο ε, λειτουργούν τα πράγματα για συνεργεία, συντήρηση, επισκευές. Θα δούμε το repair, maintenance, ε, release θα πρέπει να είναι το ίδιο ή όχι όσον αφορά και τις απαιτήσει για άλλα οχήματα. Θα δούμε το θέμα αυτό και θα έχουμε κοινή πληροφόρηση. Κύριε Παντσέρη, έχετε τον λόγο τώρα. Θα λάβετε τον λόγο για ένα τελικό σχόλιο. Παρακαλώ. Ε, Δύο λόγια μόνο κύριε Πρόεδρε. Είμαι σύμφωνος με όσα διαμειφθήκαν. Αυτό που βρίσκω σημαντικό είναι αμέσως μετά από τις 12 Απριλίου, την ε, ακρόαση δηλαδή, να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους σκιωδησηγητές όταν θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, προθεσμίες, ασφαλώς θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Επαφίεμαι στην κρίση σας κύριε Πρόεδρε και βέβαια και για τα δίκυκλα οχήματα, όπως είπατε προηγουμένως, θα δούμε τι θα προκύψει από την συζήτηση. Είναι σημαντικό να γίνουν και έρευνες ώστε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συνένεση και εδώ αλλά και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ και έχουμε ένα χρόνο διάγραμμα για να συνεργαστούμε και με το Συμβούλιο. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνάντηση εμείς και ο κύριος Φαντεκάμς επίσης για να τα δούμε αυτά. Διότι υπάρχουν κάποια θέματα που αξίζουν να εξεταστούν. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε σε αυτό το θέμα. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο ζήτημα με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Σαλβίνη υπό την πρώτη η ιδιότητα εισηγητού από τότε που προσήλθε στην Επιτροπή μας το 2009 θα έχει τη δυνατότητα έτσι να παρέμβει ως εισηγητής. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του για την ανταπόκριση στην Ευρωπαϊκή πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την προσέγγιση για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Έχετε τον λόγο κύριε Σαλβίνη να παρουσιάσετε την πρότασή σας. Έχουμε σκιώδης ο κύριος Ζουβά παρίσταται, η κυρία Γκέπαρτ παρίσταται και εκείνη, ο κύριος Κρότσμαν επίσης, Άγκστρομ επίση, εγώ, ο κύριο Τενταφυλλίδης επίσης, όλοι οι σκιώδει. Μα πιέζει βέβαια ο χρόνο κάπω, αλλά μια και υπάρχει πλήρη σύνθεση σκιωδών, υπάρχει ενδιαφέρον τουλάχιστον να έχουμε κάποια λεπτά ο καθένα για να παρέμβουμε και να συνεισφέρουμε στη δική σα σημαντική γνωμοδότηση. Κύριε Σαλβίνη, παρουσιάστε παρακαλώ το θέμα σα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τη γραμματεία της κοινοβουλευτική μας επιτροπής για αυτή τη συνεργασία. Το κείμενο είναι σχετικά σύντομο στη μορφή που πήρε για τους λόγους ή για τα στοιχεία τα οποία καθόρισαν την θέση του Κοινοβουλίου. Πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ προστασίας του καταναλωτή, που είναι το πιο σημαντικό για μας ως θέμα, και των θεμητών συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με την αντιμετώπιση των δαπανών ε, και του κόστους που έπρεπε και αυτό να ληφθεί υπόψη. Πρόκειται λοιπόν για μια συνολική προσέγγιση της προστασίας των ατόμων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε <clears throat> διασκεπτικά έξι εδάφια. Θέλαμε να διατυπώσουμε ένα κείμενο το οποίο στο μέτρο του εφικτού θα υποστηριχθεί από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και πρέπει να διαβιβαστεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών. Προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε μια ισορροπία με ένα ισορροπημένο κείμενο, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ε, και του ε, ηλεκτρονικού δικτύου και την πλατφόρμα αυτή που μυριάδες πολίτες έχουν τα στοιχεία τους και διατίθενται σε, μέσω αυτής της πλατφόρμας. Θα πρέπει να υπάρξει ένα αρμονισμός της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και εμεί από πλευράς της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας είμαστε κανονικά κατά αυτού του εναρμονισμού. Είμαστε θα έλεγα αλλεργικοί κατά του εναρμονισμού. Όμως εδώ σε σχέση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να δούμε τα θέματα προστασίας ε, των ε, προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών και τα θέματα εναρμονισμού. Επ' αυτού του σημείου λοιπόν είμαστε ανοιχτοί έναντι των διαφορετικών προτάσεων. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η Πέμπτη, 12 το μεσημέρι. Έχουμε σχετικά λίγο χρόνο. Προσπαθήσαμε όμως η προστασία των καταναλωτών να βρίσκεται στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή. Προσπαθήσαμε να δούμε ποια μέτρα για την ευαισθητοποίηση μπορούν να υιοθετηθούν και εναλλακτικέ λύσεις να αναζητηθούν και να συμπεριληφθούν. Και μια αξιολόγηση επίσης ζητήθηκε να συνταχθεί. Μια μελέτη επιπτώσεων όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πρόταση είναι ένα σχέδιο όπως είπα γνωμοδότησης ελπίζω οι παρεμβάσεις των σκιωδών να εμπλουτίσουν αυτή τη δική μου γνωμοδότηση και εσείς ο ίδιος ε, θα έχετε κάποιες ε, προτάσεις να υποβάλλετε το κείμενο είναι πολύ σύντομο όπως προανέφερα επαρκούμε σε αυτά τα σχόλια χαίρομαι για τις παρατηρήσεις σας Σας Let's Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί του θέματος αυτού, το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζει δύο νέους προβληματισμούς. Αφενός τις τεχνολογικές εξελίξεις και την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή με διαφορετικό τρόπο γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών, τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα, οι διαφημίσεις επιγραμμικώς και μετά έχουμε και την συλλογή δεδομένων, επιγραμμικά πάλι. Πώς να προστατευτούν τώρα τα προσωπικά δεδομένα. Στην έκθεση θα πρέπει να περιληφθούν θέματα σχετικά. Επίσης η ε, διαφήμιση που είναι κομμένη και ραμμένη στις επιθυμίες του καθενός, ο γεωεντοπισμός και ούτω καθεξής. Εάν δεν αναρμονίζουμε ούτε και σε αυτά τα θέματα, τότε δεν θα αναρμονίσουμε πλέον τίποτε, διότι εδώ προ, προφανώς δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το τρίτο σχόλιο έχει σχέση με τον σεβασμό των κανόνων. Νομίζω ότι η αυτορύθμιση έχει φτάσει σε κάποια όρια σε ό,τι αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν αρκεί πλέον η αυτορύθμιση, η αυτόβουλη, η οικειοθελής ρύθμιση. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι τα συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για λόγους προφανής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελεύθερης κυκλοφορίας. Ένα πέμπτο σχόλιο, η ανάγκη διευκρίνησης των συστημάτων προειδοποίησης για την παραβίαση κανόνων προστασίας δεδομένων. Όση εναρμόνιση και να κάνουμε, εάν δεν υπάρχει ένα ομογενοποιημένο σύστημα κοινοποίησης των παραβιάσεων, πάλι ε, ε, ε, φτάνουμε σε κάποια όρια. Τώρα, για το τεχνικό θέμα. προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε αυτή τη λεγόμενη privacy by design που είχε αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης έκθεσης και νομίζω ότι θα μπορέσει να αναφερθεί και στην παρούσα έκθεση. Βεβαίως τα θέματα είναι πολύ άριθμα. Συνολικά πάντως η ανάγκη παρακολούθησης των τρόπων συλλογής προσωπικών δεδομένων που δεν καλύπτονται πλέον από προηγούμενες οδηγίες, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζουβά. Η κυρία Γκέπχαρτ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαλβίνη και εσάς για την πραγματικά πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά έχει μια καλή ανακοίνωση που μας έχει υποβάλει όπου πραγματικά τα θέματα εξετάζονται τα οποία έχουν και μεγάλη σημασία. Διότι ο τομέα των προσωπικών δεδομένων και τη προστασία του είναι ένα τομέα που επί μεγάλο χρονικό διάστημα διαδραμάτισε έναν πολύ σημαντικό ρόλο για όλους στον συσχετισμό των πολιτών και του κράτους, δηλαδή των κρατικών αρχών. Κατά τα τελευταία χρόνια ή δεκαετίες έχουν αλλάξει κάποια θέματα θεμελιώδη. Η ενιαία εσωτερική αγορά, ο ρόλος της οικονομίας συνολικά σε αυτό το πλαίσιο πήρε τεράστιες διαστάσεις. Αυξήθηκε σε πολύ σημαντικό βαθμό. Είναι πραγματικά αναγκαίο να σκεφτούμε και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα τώρα πια των προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι μόνο τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ίντερνετ, μέσω ε, του διαδικτύου, ούτε των πλατφορμών Twitter, Facebook και τα λοιπά, όπου πάρα πολλά νέα άτομα δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτές τις πλατφόρμες. Πρόκειται και για το εμπόριο και για τις πάρα πολύ μικρές, ας το πω έτσι, κάρτες, ε, ε, δελτία, πληροφορίες και στοιχεία, όπου οι πολίτες τις επιθυμίες ή την εικόνα ε, για την αγορά ενός προϊόντος και τα χαρακτηριστικά δίνουν. Πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες για να γνωρίζουν οι πολίτες τι θα κάνουν σε σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ ευρύ φάσμα λοιπόν, ευρύτατο φάσμα που πρέπει να καλυφθεί από εμά εδώ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρόκειται πραγματικά εδώ όχι μόνο για δικαιώματα των πολιτών, αλλά και για θέματα της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και για θέματα προστασίας των καταναλωτών. Πολύ περισσότερα αυτά στη γνωμοδότηση πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το ξέρω κύριε Σαλβίνη, πάντα έχουμε πολύ λίγο χώρο για τις γνωμοδοτήσεις και κάποια πράγματα πρέπει να παραμένουν εκτός. Όμως Αυτά πρέπει να τα εντάξουμε θα έλεγα. Πρέπει να θέσουμε ιδιαίτερη έμφαση και εσείς το έχετε στην γνωμοδότησή σας με ιδιαίτερη έμφαση να αναφερθούμε στο πώς, πώς η διαφάνεια στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων θα εισαχθεί. Πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε και για κάτι άλλο, να υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης αυτών των στοιχείων, ανάκτησης και ανάκλησης και το δικαίωμα για, στην επιστροφή στοιχείων ή ακύρωσης να ενισχυθεί δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας, η προστασία της ιδιωτικής ζωής ε, μέσω αυτών των πράξεων. Έχουμε μια σωστή βάση που μπορούμε να την ενισχύσουμε και θα καταθέσω κι εγώ αντίστοιχες τροπολογίες γι' αυτό. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέφαρτ. Ο κύριος Κρόιτσμαν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίως να συγχαρώ τον συνάδελφο Σαλβίνη για, αυτή την πάρα πολύ, για αυτές τις πολύ καλές προτάσεις που υποβάλλει. Επειδή είναι περιεκτικές και περιεκτικά με συμπυκνωμένο τρόπο λαμβάνουν υπόψη τα προβλήματα και τα καλύπτουν για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πρώτον, για τους νέους ιδιαίτερα η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική, μια και οι νέοι είναι πολύ γενναιόδοροι στη διάθεση αυτών των προσωπικών δεδομένων τους. Και έτσι η διαγραφή, η ανάκληση των προσωπικών δεδομένων που αναφέρεται στη δική σας νομοδότηση πολλές φορές ε, ε, ε, αντιμετωπίζει προβλήματα και πρέπει να μεριμνήσουμε να καταλήξουμε σε σωστές λύσεις. Δεύτερον, η οικονομία πρέπει να γνωρίζει ποια στοιχεία προσωπικά θα μπορούν να αποθηκεύονται και ποια όχι. Γι' αυτό ένας εναρμονισμός, και εσείς το αναφέρετε αυτό ρητά, στο ευρωπαϊκό επίπεδο εναρμονισμός είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Βοηθάει αυτό να αναπτυχθεί ένα τμήμα ακόμα παραπέρα τη ενιαία εσωτερική αγορά. όταν θα έχουμε κοινέ προδιαγραφέ για τι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Και τρίτον, και αυτό θέλω να το τονίσω, χαιρετίζουμε ότι η επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, Διότι εξαρτώνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσει τα κόστη τα οποία θα επιβάλλονται σε αυτές και θα τις επιβαρύνουν να είναι μικρά, μικρότερο, μικρότερα αν γίνεται γιατί είναι δυσανάλογα σήμερα και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Γι' αυτό η επιβάρυνση των ΜΜΕ πρέπει να είναι, μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να είναι λογική. Συνολικά είναι πολύ καλές αυτές οι προτάσεις, τις υποστηρίζουμε και θα δούμε αν με τροπολογίες μπορούν να συμπληρωθούν. Ευχαριστούμε. Ε, Mr. Engstrom. Συμφωνώ με τους προηγούμενους. Η γνωμοδότηση είναι καλή. Και το έγγραφο εργασίας της ΛΥΜΠΕ επίσης είναι επαρκές. Όντως χρειάζεται νομοθεσία εν προκειμένου διότι δεν αρκεί η λεγόμενη αυτορύθμιση. Και σωστό είναι επίσης να γίνει η νομοθεσία αυτή στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υπάρχουν και ίσοι όροι ανταγωνισμού για να μπορούν να εργάζονται και διαμεθοριακά οι διάφορες επιχειρήσεις. Όπως είπα λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Ταυτόχρονα δεν θέλουμε να είναι και υπερβολική η νομοθέτηση αυτή, γιατί είναι εύκολο να ξεπεράσει κανείς κάποια όρια. Υπάρχει νομοθεσία αυτή βέβαια από τη δεκαετία του 70. Κάποια στιγμή υπήρξε στην Σουηδία μια περίπτωση όπου κάποιος έγραψε κάτι σε ένα blog, κάτι λίγο ε, ε, εκτός όριων για κάποιους φίλους και δυστυχώς όπως είναι οι κανόνες στην Σουηδία μπήκε στο πεδίο εφαρμογής του νόμου διότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε σχέση με ιατρικό απόρριτο για το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο ήταν θέμα υγείας δηλαδή, ε, και εκεί βέβαια βρέθηκε ε, απέναντι σε σημαντικέ δυσκολίε. Τώρα, το να λησμονηθούν τα δεδομένα, εγώ δεν ξέρω ακριβώ τι σημαίνει. Εάν σημαίνει ότι εάν αποχωρήσω από το Facebook, το Facebook θα πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα, αυτό είναι σωστό. Και ε, αυτό θα πρέπει να προβλέπουν και οι κανόνες. Από την άλλη μεριά, εάν σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να σε ξεχάσουν. Ε, ε, ένα παράδειγμα, ορισμένοι πρώην ευρωβουλευτές θα ήθελαν να ξεχάσει ολόκληρο το διαδίκτυο ότι ήταν διατεθειμένοι κάποια στιγμή να πουλήσουν τροπολογίες για χρήματα, δηλαδή να ε, εισπράξουν χρήματα για να προβάλλουν τροπολογίες. Αυτό ίσως θα έπρεπε να μπορεί να γίνει, από την άλλη μεριά δεν θα ήταν και κατάλληλο, αν είναι δυνατόν δηλαδή, να διαγραφούν πράγματα ε, για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο ε, που έχουν πει άλλοι. Τέλος πάντων, χρειάζεται να εξευρεθεί μια λεπτή ισορροπία αλλά γενικά το κείμενο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ εν τέλει, ευχαριστώ εν τέλει τον εισηγητή. Uh, uh Mr. Κύριε Τριανταφυλλίδη, παρακαλώ. Thank you, Chairman, and uh, many thanks to... Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τον κύριο Σαλβίνη για την ε, θαυμάσια δουλειά. Η... Ο σεβασμός της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και των προσωπικών δεδομένων είναι και θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βέβαια, είναι και δύσκολο να διατηρηθούν τα δικαιώματα αυτά μέσα σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο ψηφιακό κόσμο, όπου σημειώνεται τέτοια ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και γι' αυτό πρέπει να είναι εξασφαλισμένο ώστε στη μελλοντική νομοθεσία να παραμένουμε τεχνολογικά ουδέτεροι, ώστε η προστασία να ισχύει ούτω ή άλλω, ανεξάρτητα δηλαδή από την τεχνολογία συλλογή των δεδομένων και κανένα χώρο να μην αποκλείεται από την προστασία, από τους, από τους κανόνες προστασίας. Οι διατάξει λοιπόν προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να καλύπτουν από τους καταναλωτές online μέχρι και τους ε, εργαζομένους σε σχέση με τους εργοδότες και ούτω καθεξής. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί είναι μέσω της ομοιογενειοποίησης ομογενοποίησης των ε, ε, εθνικών νομοθεσιών, γιατί έχουμε δει τα τελευταία 15 χρόνια πολλές μεγάλες αποκλίσεις στις νομοθετικές διατάξεις των χωρών μελών. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και περισσότερο, δηλαδή να προβλέψουμε ενιαίους ορισμούς για την συλλογή των ε, προσωπικών δεδομένων, την επεξεργασία τους, τις διεθνείς διαβιβάσεις τέτοιων δεδομένων τις ε, αρχές εποπτείας και ούτω καθεξής. Και όπου δεν γίνεται επισήμως η συλλογή δεδομένων σε ευρωπαϊκό έδαφος, το λεγόμενο cloud computing. Εν τέλει, κύριε Πρόεδρε, η συνειδητοποίηση του κοινού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε όλες τις χώρες μέλη. Και αυτό μπορεί να γίνει εάν ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Αλλά όχι μόνο. Η συνειδητοποίηση θα πρέπει να γίνει και με ενημέρωση των ατόμων σχετικά με την ανάγκη προστασία των, προστασίας των δεδομένων τους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ως κοιόδηση ο θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση ε, σωστά ο κ. Σαλβίνη εστιάζει ε, στη διάσταση της ενίας αγοράς. Στην έκθεση της Κομισιόν υπάρχει και συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε κάποια από τα θέματα που αναφέρει αυτό το κεφάλαιο στην στο κείμενο της Κομισιόν. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προσπαθεί να δει σε ποιο επίπεδο θα γίνει η εναρμόνιση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων. Όπως λέει και παραθέτω, η οδηγία μερικές φορές έχει εφαρμοστεί ε, όχι με σωστό τρόπο από τα κράτη-μέλη. Αυτό ε, είναι πρόβλημα της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, διαστάσεις μεταξύ των εθνικών κανόνων και των οδηγιών και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Η Κομισιόν πρότεινε κάτι εντελώ καινούριο, δεν το κατάλαβε εντελώ. Ε, Πάντω, ούτω ή άλλω, οι ισχύοντε κανόνε θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά, με συνεκτικό τρόπο. Σωστά, επίση, ε, εντοπίζει κάποια θέματα που αφορούν την κοινοποίηση. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι εδώ που θα πρέπει να ενισχυθεί στην έκθεση Σαλβίνη. Υπάρχει συνένεση μεταξύ των ελεκτικών αρχών ότι η σημερινή υποχρέωση να κοινοποιήσουμε ε, είναι μια επαχθής διαδικασία που δεν δίνει προστιθέμενη αξία για την προστασία, σε ό,τι αφορά την προστασία των ατόμων. Υπάρχει λοιπόν ε, συνένεση μεταξύ των ελεκτών για την προστασία των δεδομένων ότι θα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτό, ε, ούτω ώστε να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η μείωση του διοικητικού άχθους αλλά και η βελτίωση της προστασίας των δεδομένων. Η πρόταση επίσης να ενισχύσουμε το ρόλο του, της ομάδας εργασίας 29, που είναι η ομάδα εργασίας όπου οι ελεγκτές προστασίας των δεδομένων συνέρχονται για να συντονίζουν τις δραστηριότητε τους και να αποκτήσουν έτσι πιο θεσμοθετημένο ρόλο, ε, εφαρμόζοντας τους τυποποιημένους κανόνες, παρά να, να υποστηρίξουμε ένα σώμα όπως ανάλογο αυτό ε, όπως ανάλογο με τους ελεγκτές για τις επικοινωνίες, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για να σημειώσουμε πρόοδο. Κάτι άλλο τώρα. Για την ε, παραβίαση της υποχρέωσης κοινοποίησης ε, των προσωπικών δεδομένων. Ως εισηγητή σας, αγαπητοί συνάδελφοι, για τα δικαιώματα των χρηστών ε, στο πακέτο μεταρρύθμισης για τις τηλεπικοινωνίες, θα θυμάστε ότι συνεργαστήκαμε πολύ στενά με την Επιτροπή Αστικών Ελευθεριών για τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για την ιδιωτική σφαίρα, που ήταν και ενέρη ευθύνη μας και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο για την κοινοποίηση παραβίαση των προσωπικών δεδομένων που ισχύει αυτή τη στιγμή για τις ε, εταιρείε τηλεπικοινωνιών. Ο κ. Σαλβίνη λέει ότι αυτή είναι μια πρόταση ε, επαχθής και ε, ακριβή. Οι νέε προποθέσει ακόμα δεν έχουν ισχύσει και κάναμε μεγάλη προσπάθεια με τι ελληνικέ αρχέ, ούτω ώστε να μην είναι αυτή η πρόταση ούτε επαχθή ούτε ακριβή στην εφαρμογή. Και χαίρομαι που το έργο που έκανε η Επιτροπή μας περνάει σε όλους τους κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Έγκστρομ, σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αυτό το δικαίωμα να ξεχαστείς πρέπει να, το, να ξεκινήσει από σένα. Ό,τι έχουν γράψει άλλοι για σένα είναι και στον κυβερνοχώρο και δεν έχει κανέναν έλεγχο για αυτό το θέμα. Έτσι, νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι βάζουν διάφορα στοιχεία στο facebook ε, όταν είναι νεαροί και μετά το μετανιώνουν όταν είναι πιο μεγάλοι και όριμοι. Αλλά αυτό πρέπει να μπορούμε λοιπόν να το ρυθμίσουμε. Αυτά κύριε Σαλβίνη. Η κυρία Μπουλανζέ που είναι επικεφαλής τομέα στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης είναι εδώ μαζί μας, θα μας κάνει λίγα σχόλια και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαλβίνη. Κύριε Μπουλανζέ, μπορείτε να κάνετε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε μεγάλο ενδιαφέρον την σημερινή συζήτηση και τα επιμέρους ε, σημεία που συμπίπτουν με τα σημεία που εξέτασε η Κομισιόν από πλευρά τη, στα πλαίσια προετοιμασίας μιας ανάλυσης αντικτύπου εν ώψη μια νομοθετική που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή κέρι. Για να δούμε αν τελικά θα προτείνουμε νομοθετικό κείμενο ή και για να, πάρουμε υπόψη μας, να λάβουμε υπόψη μας και τα τελευταία σημεία που ακούσαμε. Η διάσταση για την εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντική για μας. Είναι από τα σημεία τα οποία εντοπίσαμε ως μία από τις αδυναμίες του σημερινού συστήματος και στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε για την περαιτέρω αναρμόνιση δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε περιττό γραφειοκρατικό άχθος, δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ που πήρατε την πρωτοβουλία για αυτήν την πρόταση, ε, την οποία μας, είχε, μας υποσχέθηκε η κυρία Ρέντιν πριν ε, από τις εκλογές. Ε, χαίρομαι λοιπόν που ανταποκρίνεται η κυρία Ρέντινγκ, ε, ιδίως για το θέμα της ε, κοινοποίησης παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Μέχρι τις 12 η ώρα την Πέμπτη έχετε ε, την ε, δυνατότητα να υποβάλει τροπολογίε. 12 Απριλίου θα εξετάσουμε τι Απριλίε. 25 και 26 Μαΐου θα ψηφίσει η Επιτροπή Αστικών Ελευθεριών και θα ψηφίσει η Ολομέλεια τον Ιούνιο. Κυρία Σαλβίνη, θέλετε να συνοψίσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ τους έξι ομιλητές που πήραν τον λόγο. Θέλω να καθησυχάσω τον κύριο Ζουβά για το επίπεδο εναρμόνισης. Ε, το επίπεδο εναρμόνισης, κατά την αποψή μας, θα πρέπει να είναι το μέγιστο δυνατό. Όπως είπε και ο κ. Τριανταφυλλίδη, τα δεδομένα που συλλέγονται στις 27 χώρες μπορούν να φτάσουν στα πέρατα του κόσμου. Επομένως, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όποιος συλλέγει είναι ε, πρέπει να ξέρει σε ποιον θα δίνει τα δεδομένα, ε, πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες ε, και στα 27 κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία σε αυτό. Επίσης θα πρέπει αυτό να επισύρει το λιγότερο ε, άχθος, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που καμιά φορά η συλλογή δεδομένων αποτελεί τρομακτικό βάρος. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα, να εξασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία. Ε, για, την, για που είπε ο κύριος Κρόιτσμαν και η κυρία Γκέπχαρτ, ε, για τη δυνατότητα ανάκλησης, αν θέλετε, των δεδομένων. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για το πώς, ε, τι επεξεργασία υφίστανται τα δεδομένα τους και μέσα από, ποιες, ε, μέσα από ποιους διάβλους ας πούμε τα δίδονται. Γιατί εγώ μπορώ ας να είμαι στο facebook, θα πρέπει να ξέρω τα δεδομένα μου, ε, ποιοι άλλοι κοινωνικοί εταίροι, ποιοι άλλοι χρήστες τα χρησιμοποιούν, πού αλλού μεταδίδονται. Ε, το δικαίωμα λήφθης. Εδώ είναι μία άλλη συζήτηση που δεν μπορεί να ενταχθεί στην σύντομη μικρή μας συζήτηση. Είναι μεγάλο αυτό το θέμα. Το θέμα ότι θα πρέπει να υπάρχει μέγιστη δυνατή ομοιομορφία, όπως είπε ο κ. και ο κύριος Χάρμπορ, συμφωνούμε απόλυτα. Δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Ούτε χρόνο, ούτε χώρο, γιατί Είμαστε μία από τις επιτροπές που γνωμοδοτούν. Μέχρι την Πέμπτη περιμένω τις τροπολογίες σας ε, για να εξυπηρετήσουμε τα εκατομμύρια χρηστών και καταναλωτών που αυτή τη στιγμή ε, αντιμετωπίζουν διαφορετική εντελώς μεταχείριση ε, στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Σαλβίνη. Περιμένουμε λοιπόν τις τροπολογίες και την τελική συζήτηση. Πάμε στις ψηφοφορίες. Έχουμε διάφορες σημαντικές προφορίες. Πρώτα απ' όλα θα δούμε τα ονόματα για τα κλωστοϊφαντουργικά και τις ονομασίες. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μάντας. Και ενώ το κάνουμε αυτό, όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες να διασφαλίσουν ότι οι ομάδες τους θα, είναι συναθρισμένες με κάρτες ε, για την ψηφοφορία για το θέμα του κύριου Μάντας. Κύριε Μάντας, θα θέλατε να μας ε, παρουσιάστε τις τροπολογίες και αν κάποιος από τους σκιώδεις θέλει να παρέμβει, παρακαλώ. Μπορείτε να παρέμβετε, αλλά ελπίζω ότι ο κύριος Μάντας θα σας ικανοποιήσει με τις παρεμβάσεις του και έχει και προτάσεις για ομού ψηφοφορίες, από κοινού ψηφοφορίες. Έχει τον λόγο κύριε Μάντας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Φυσικά πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την πολύ αποτελεσματική συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές, διότι πραγματικά είναι καλό, θετικό να βλέπει κανείς πως όλοι παρακολουθούν τις συνεδριάσεις που προβλέπονται και διοργανώνονται και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε όπως πρέπει και να βρίσκουμε ένα γενικό συμβιβασμό προς όφελος όλων. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τις νομικές υπηρεσίες. Έκαναν εξαιρετική δουλειά για αυτά τα θέματα. Γενικά αυτά τα οποία πρόκειται, αυτά περί των οποίων πρόκειται εδώ για την, για τον πίνακα ψηφοφορίας για την πρώτη ανάγνωση και έγκριση σε πρώτη ανάγνωση έχουμε κάποιες ίσονο σημασία ε, τροποποιήσεις και αλλαγές λόγω τροπολογιών και θα ψηφιστούν αυτές ε, και με προφορικές τροποποιήσεις. Είναι μια βελτίωση του κειμένου μόνο όλο και όλο. Και για, κατά τα άλλα ελπίζω ότι μπορούμε να υπερψηφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες en bloc, ομού, από κοινού, για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί έχουμε καθυστέρηση 20 λεπτών όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά μας. Και έτσι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με την από κοινού ψηφοφορία τροπολογιών να ρυθμίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ όλους σα πολύ λοιπόν. Και για τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών αυτή τη κοινοβουλευτική επιτροπή που θα ήθελα να έχουμε ή ομόφωνη υπερψήφιση, θα μπορούμε έτσι να έχουμε μια ισχυρή θέση και τοποθέτηση για τι διαπραγματεύσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει περισσότερο, κατά το μάλλον ή τον τη γραμμή μα, και το Συμβούλιο προσπαθεί να συζητήσει κάποια θέματα και να δεχτεί κάποια, προτάσει. κάποιες προτάσεις. Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε γοργά ένα συμβιβασμό και το απόγευμα θα παρακολουθήσω τη συνάντηση των συντονιστών για να δούμε αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει τις άτυπες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το δυνατό πιο γοργά να εγκρίνουμε αυτόν τον κανονισμό. Το να υπάρξουν νέες ίνες στην αγορά είναι ένα από τα πιο σημαντικά τεχνικά θέματα ως πρόταση. Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση. Και για τα πολιτικά θέματα που θέλουμε να περάσουν ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αυτό είναι σημαντικό, μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό, ελπίζω, με το Συμβούλιο στο τέλος. Ας ψηφίσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση. Θα δούμε αν όλοι μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις προτάσεις. Να έχουμε μια ισχυρή λοιπόν θέση όσον αφορά την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο στη συνέχεια. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς θα θέλατε να παρέμβετε, κυρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μάντερς και όλους τους υπόλοιπους και όλους τους εισηγητές, γιατί αυτό το θέμα είναι δύσκολο. Και όλα αυτά είχαμε μία συνεπή θέση από την αρχή. Από το 2009 δηλαδή μέχρι τώρα και στη δεύτερη ανάγνωση ενδυναμώνουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Και αυτό πώς καθίσατε δυνατόν αν έχουμε μια ομόφωνη ψήφο. και να είμαστε πιο δυνατοί. Ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συνεργασία και ελπίζουμε ότι αυτό αυτή η ψήφος θα είναι σημαντική και καθοριστική για το Συμβούλιο. σωστά. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και θα ψηφίσουμε. Δεν χρειάζονται νομίζω θα έλεγα ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε αυτό το γύρο. Περνάμε λοιπόν στην ψήφισή τους άμεσα και ακολουθούμε τις ομού ψηφοφορίες όπως πρότεινε ο εισηγητής. Αν κάποιος θέλει κάτι διαφορετικό, αυτά έχουν συμφωνηθεί με τους κοιόδης, αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουμε. Άρθρο 1 λοιπόν, τροπολογία 10 του κυρίου Μάντερς, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα. Μετά, άρθρο 2 για το εύρος. Η κυρία Μακλάκιν, η τροπολογία της 38, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Περνάμε σε ομού ψηφοφορίες ε, του, για τροπολογίες του κυρίου Μάντες. Από το 12 στην 20, για τα άρθρα 4 και 9 και μέχρι και το 15 άρθρο. Αυτές οι τροπολογίες λοιπόν, μέχρι την 20 υπέρ, κατά εγκρίθηκαν αυτές οι τροπολογίες. Περνάμε στο μπλοκ 4 μετά στη συνέχεια. Τροπολογία 21 με την προφορική τροποποίηση που προβλέπεται στο έγγραφο μέχρι την 43 ε, τροπολογίες υπέρ. 21 έως 40 υπέρ κατά εγκρίθηκαν αυτές. Τώρα περνάμε στην ομού ψηφοφορία υπαριθμών 5. Όλες οι τροπολογίες στο άρθρο 18, 22 28, σωστό, μάλιστα, υπέρ αυτών, κατά, εγκρίθηκαν και αυτές και μετά η ομού ψηφοφορία στην ομάδα 6, μπλοκ 6, τροπολογία 41-42, όλες στο άρθρο 24α, υπέρ, κατά, εγκρίθηκαν, μετά η 43 αυτοτελώς υπέρ κατά εγκρίθηκε Περνάμε στο μπλοκ 8, τροπολογίες 31 έως 34, υπέρ αυτών. Κατά εγκρίθηκαν. Και τώρα πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Δεν έχουμε να ψηφίσουμε κάτι εκεί. Πάμε στο 9, τροπολογία 4 σχετικά, ένα συμβιβασμό. Τροπολογία 4 με την προφορική τροποποίηση υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Θα πρέπει να καταμετρηθούν οι ψήφοι. Πρέπει να καταμετρήσουμε. Εντάξει, ηλεκτρονικά. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο. Δεύτερη ανάγνωση. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 30 ψήφοι υπέρ 2 εναντίον 4 αποχές μέσα στις ποσοστώσεις όλες οι ομάδες μάλιστα εντάξει και σύμφωνα με τη μηχανή βρίσκεστε μέσα στις ποσοστώσεις των ομάδων από τον αριθμό ψηφοφόρων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάντες και θα προσέθετε στη συνάντηση των συντονιστών για την εντολή, για την ένταξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Εντάξει, προσβλέπουμε λοιπόν στη συνεργασία σας σήμερα το απόγευμα. Περνάμε στην ε, γνωμοδότηση της κυρίας Κόρολα. χαιρετίζω την Αντιπρόεδρο για το εύρος ε, των ε, του ραδιοφάσματος. Θα σας δώσω τον λόγο για να μας παρουσιάσετε τις τροπολογίες παρακαλώ. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μαζί και για την ελαστικότητα που κατέδειξαν στην προσέγγιση αυτών των τροπολογιών. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την υπομονή που κατέδειξε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με τους συμβιβασμούς και τα αποτελέσματα που επετέφθησαν και ελπίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια σωστή ισορροπία και ένα πολλά υποσχόμενο αποτέλεσμα. Δεν έχω άλλα σχόλια, ας ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κάποιος Γιώδης θα ήθελε να σχολιάσει. Όχι, ξεκινάμε με τις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε το άρθρο 1. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίθηκε. Δεν θα ψηφίσουμε την 52. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογίες 54 και 55 υπέρ αυτών κατά εγκρίθηκαν. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό 1 υπέρ κατά Α, σαφώς εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στο 9 σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Κορόλα υπέρ θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. DO9 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 24 υπέρ 12 εναντίον. Η τροπολογία 59 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίθηκε. Η τροπολογία 60 Κρόιτσμαν υπέρ κατά και αυτή εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στον συμβιβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε σαφω. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 63 και 64 που είναι ταυτόσιμε οι δύο του. 63 και 64. Υπέρ αυτών. Θα αρχίσει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά όμω. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 63 και 64. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα ψηφοφορία. Απορρίφθηκαν. 21 ψήφος, 21 ε, ψήφοι εναντίον, 15 ε, υπέρ, 65 τροπολογία, Μπομπίνσκα υπέρ, κατά, εγκρίθηκε και μετά τροπολογία 66, Μπομπίνσκα υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Στη συνέχεια για το άρθρο 4 έχουμε δύο ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ αυτών, κατά, εγκρίθηκαν, τροπολογία 68, Κρόισμαν υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 69, de Μόζε, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Το σχέδιο 12 καταπίπτει, τροπολογία 70, Μπομπίνσκα, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 71. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε την 71 τροπολογία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 72, Hans Peter Mayer, υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 72. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 25 ψήφοι υπέρ 11 εναντίον. Και περνάμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 73, Μπομπίνσκα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 74, Μπομπίνσκα, υπέρ, κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 76 και τροπολογία 77 από κοινού είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε 76 και 77. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Τροπολογία 75, Hans Peter Mayer, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Μετά περνάμε στις τροπολογίες 78, 79 και 80. Από κοινού με την προφορική τροποποίηση που προτείνεται υπέρ, κατά, εγκρίθηκαν. Και έτσι οι κύριες τροπολογίες ε, σχετικά καταπίπτουν. Περνάμε στο συμβασμό 3, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στη συνέχεια στο σχέδιο 15 της κυρίας Κόρολα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το 15 της πρότασης Κόρολα. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 19 ψήφους υπέρ 14 εναντίον και έτσι οι 88, 89, 90 καταπίπτουν, 91 Κρόισμαν υπέρ κατά εγκρίνεται. 92 καταπίπτει. 92-93 καταπίπτουν. Τροπολογία 94. Μπομπίνσκα υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε σαφώς. Η τροπολογία 95 αρκετό συναδέφων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 95. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 20 ψήφοι υπέρ 16 εναντίον. Τροπολογία 96. Έγκερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 96. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Η 97 καταπίπτει. Η 216 καταπίπτει. Περνάμε 217 κόρολα υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το 17 της ε, γνωμοδότησης κυρίας Κόρολα. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Περνάμε στην 98 κόρολα. Σωστό. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 98. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, η 2.18 καταπίπτει τροπολογία 99, Μπομπίνσκα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 99 Μπομπίνσκα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε αυτή. Και περνάμε στο άρθρο 8. Τροπολογία 19 Κόρολα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το 19 Κόρολα. Πέρα, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Οι τροπολογίες 100 και 101 καταπίπτουν. Θα ψηφίσουμε τα 102 και 103 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ αυτών, κατά, εγκρίθηκαν. Το 220 20 ως προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία για το 20. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Η 104, Μπομπίνσκα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τώρα για το άρθρο 9. Τροπολογία 105. Σαν Μόζερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 105. Τέλος ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε την 21 κόρολα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 21. Τέλος ψηφοφορίας. Σαφώς εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 24. Μπομπίνσκα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2-2. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 2-2 της κυρίας Κόρολα. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 25, Μπομπίνσκα. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 26, Γκρέκ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η τρία της κυρίας Κορόλα, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε τη τρία Κορόλα. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. Και έτσι η τροπολογία 27 είναι προσθήκη σε αυτό. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 κόρολα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 28 και 29. Ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτών. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Τροπολογία 31 Κρόισμαν υπέρ, κατά, α, εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 Hans Peter Mayer υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 30 ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίθηκε η 30. Τροπολογία 32, Μπομπίντσκα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 33 Μπομπίνσκα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 34 Hans Peter Mayer. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε σαφώς. Το 25 εγκρίθηκε, καλύπτεται. Η τροπολογία 35 θα ψηφίσουμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 35. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά εγκρίθηκε και περνάμε στη συνέχεια στο τέλος μέχρι την τροπολογία συμβιβαστική τροπολογία 6 πρώτα ναι, συμβιβαστική 6 υπέρ της συμβιβαστικής 6 κατά εγκρίθηκε και τώρα πάμε στην τροπολογία 47, Σάλντε Mose. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 47. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία... Α, 46. Όχι, 48, συγγνώμη. Πρόεδρος 48, Κόρισμαν υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 49 και 50, υπέρ αυτό Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε 49 και 50 ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκαν. Και τώρα θα ψηφίσουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολό του, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης στο σύνολο. Τέλος ψηφοφορίας ένας αποφάσισε να μην ψηφίσει για την νομοδοσία σας ε, και εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ και μία ψήφο εναντίον. Συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή τη δουλειά που κάνατε. So I'd like to thank Mrs. very much. Ευχαριστώ την κυρία Κορόλα για το σημαντικό της κείμενο. Θα υπερασπιστώ τις τροπολογίες μας στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Θα ψηφίσουν σύντομα εκεί στις 12 Απριλίου, αν δεν απαντώμε. Και εν συνεχεία θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Και τώρα περνάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης για το Ευρωπαϊκό Εταιρικό, ε, μάλλον συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ε, Συμβάσεων. Hans Peter Mayer. Υπάρχουν ε, μία-δύο προφορικές τροπολογίες που θα πρέπει να σταθούμε. Ο κύριος Μάγερ είναι εδώ. Όχι, δεν είναι. Ο κύριος Βάπ τον αντικαθιστά. Θέλει να πει κάποια εισαγωγικά πράγματα. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε δεν είμαι ο ίδιος εισηγητής της νομοδοτήσεως αυτής της Νομικής Επιτροπής αλλά ο κύριος Μάιερ ασθενής σήμερα όπως και χθε. Θα κάνω δύο σύντομα σχόλια πριν αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Πρώτα, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι εν τέλει η λίστα ψηφοφορίας διαβιβάστηκε με καθυστέρηση στους συναδέλφους. Δεν ε, με βαρύνει το κρίμα αυτό, αλλά εκφράζω τη λύπη μου παρόλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει κάποιες περιστάσεις και ευθύνη πολλών οδήγησαν σε αυτή την καθυστέρηση. Δεύτερο, χθε είπαμε ότι έχουμε μια συμβιβαστική πρόταση για τις 24, 27 και 56 τροπολογίες που τις συγχωνεύει αυτές σε ό,τι αφορά τη μελέτη επιπτώσεων οφείλουν να εξεταστούν όλες οι επιλογές σε σχέση με τις πραγματικές επιπτώσεις, το κόστος και τις υφιστάμενες επιλογές. Επίσης, η νομική βάση, οι κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις, οι διασυνδέσεις με το εθνικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, με δίκαια επιλύσεως διαφορών, μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να εξεταστούν. Μια ολόκληρη σειρά συνθήκων δηλαδή που είναι απαραίτητες για την εξέταση των επιλογών και για την 56 τροπολογία πρέπει να ληφθεί υπόψη για παράδειγμα και η οδηγία προστασίας των καταναλωτών. Μπορώ να επεκταθώ περισσότερο, αλλά θέλω με λίγα λόγια να πω ότι μέσα στον συμβασμό περιλάβαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να συνεξεταστούν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να συμφωνήσουν οι συνάδελφοί μου. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις ηγητές θέλουν να σχολιάσουν. Όχι. Ας ψηφίσουμε. Θα είμαι πιο αργός, γιατί υπάρχουν κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Επίσης υπάρχει και μία συμβαστική προφορική τροπολογία που θα δούμε σε λίγο. Πάμε στην παράγραφο 1 Τροπολογία 24. Από διάφορους συναδέλφους. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25 καταπίπτει τότε. 26 και 29 ψηφίζουμε μαζί. Είναι ίδιες τροπολογίες. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο. Η κυρία Ρούλε ε, με την τροπολογία της 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 89. Τον κύριο Κρέχα. Υπέρ. Ναι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 89. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 16... 18 κατά, 16 υπέρ. Τροπολογία 28. Ζουβέν και τα λοιπά. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώ. πάμε στην παράγραφο 2 τώρα. Έχουμε μια αποφορική τροπολογία εδώ, που είναι συμβιβαστική. Ε, σοσιαλιστές, ε, συντηρητικοί μαθητιστές, αριστεροί και η Ευρώπη των, ε, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Θα ήθελα Καταρχά, υποθέτω ότι θέλετε να ψηφίσετε την προφορική τροπολογία. Ναι, θέλετε. Μια και είναι η πιο ρηξικέλευθη, θα πρέπει να την ψηφίσουμε πρώτα. Και αν καταπέσει, θα ψηφίσουμε το συμβασμό. Συμφωνείτε. Ο κύριος Φάμπ. Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα λίγο την κατάσταση και οι δύο Αυτές οι τροπολογίες κατατέθηκαν μετά από την προθεσμία, τη λήξη της προθεσμίας. Έχω λοιπόν διαδικαστικά την εντύπωση ότι μπορούμε να ψηφίσουμε μόνο την συμβαστική τροπολογία, ή μάλλον πρώτη τη συμβαστική τροπολογία του εισηγητού. Δεν έχω βέβαια πραγματικά μελετήσει σε βάθος ώστε να αποκλείσω όλα τα ενδεχόμενα, ίσως μπορεί η μαλλον πρωτη τη συμβαστικη τροπολογια του εισηγητου δεν εχω βεβαια πραγματικα μελετησει σε βαθος ωστε να αποκλεισω ολα τα ενδεχομενα μπορει η γραμματεια να μας φωτίσει. Είναι περίπλοκο το θέμα. Μάλλον θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη συμβαστική τροπολογία. Μια και πρόκειται όμως για συμβαστικές τροπολογίες, θα πρέπει ο πρόεδρος να αποφασίσει. Και κατά την άποψή μου, η... αυτή η τροπολογία των σοσιαλιστών είναι πιο μακριά από το κείμενο. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το συμβασμό πρώτο. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία των σοσιαλιστών, ECR, GUE, και η με ονομαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν τον πρώτο συμβασμό. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δίσταζα. Γιατί δεν ήξερα αν είμαστε όντως 36, όχι μάλλον είμαστε 36, 20 ε, κατά, 16 υπέρ, απορρίπτεται. Πάμε τώρα το, να ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία 1. Έτσι. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με 20 ψήφους υπέρ και 15 κατά. Τότε πάμε κατευθείαν στην ε, τροπολογία 34, αν δεν απατώμε. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί λέμε εδώ πέρα ψήφο κατά τμήματα. Τι χωρίζουμε εδώ πέρα. Το δεύτερο τμήμα. Α. Υπέρ του δεύτερου τμήματος κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 37 του Λουί Γκρέχ. Ένα προφορίας για την 37. Πέρας. εγκρίνεται. 22 υπέρ, 14 κατά, 38 του ιδίου υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε 38. Ένα ψηφοφορίας, πέρας. Εγκρίνεται επίσης. 39. Στάιλερ. Ξεκινάμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 39. Πέρας. Καταπίπτει. Έχουμε ακριβώ τον ίδιο αριθμό ψήφων. Σωστό δεν είναι αυτό που λέω. Ναι, λίγο γραμματέ. Πάμε στην ε, τροπολογία 40 του κ. Φόξ. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται σαφώς. 41. Μακλάκιν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται σαφώς. 42. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι η 43 καταπίπτει. Πάμε στον συμβασμό υπαριθμών 2. Πάμε στον δεύτερο συμβιβασμό, υπέρ. Θα ψηφίσουμε φωνικά καλύτερα για την δεύτερη συμβαστική τροπολογία. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τότε πάμε στην τροπολογία 49. Ξεκινάει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Επίσης απορρίπτεται. 52 και 53 μαζί. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε την 54. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 56. Σμιτ. Νέα παράγραφος. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57 και 60 ψηφίζουμε μαζί. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Ίδιο αριθμό ψήφων και εδώ καταπίπτει λοιπόν. 59. Έναξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 63. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ε, έχουμε τώρα την 61 και 65, που είναι ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας για το πρώτο τμήμα της 61 και 65. Πέρας. Εγκρίνεται. Τότε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Όπως βλέπετε στο κατάλογό σας, ξεκινάμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά στο δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο υπέρ διαφορά. Τώρα είμαστε 35 αυτοί που ψηφίζουν. Με μυστηριώδη τρόπο δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί μειωθήκαμε. Πού πάμε τώρα. Πάμε στην 62. Εμεί θεωρούμε ότι ψηφίζουμε τώρα την 62. Συμφωνείτε? Ωραία. Ξεκινάμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία. Α, πάλι ψηφίσαν 36. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την 61 και 65, το τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Περνάει σαφώς. Παράγραφος 9 τώρα. Πάμε στην παράγραφο 9. 67 και 70 μαζί. Τις ψηφίζουμε, έτσι, αυτές τις δύο. Υπέρ, παρακαλώ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Την 67 και 70. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όλες οι άλλες τροπολογίες αυτής παραγράφου καταπίπτουν και πάμε στην ε, συμβαστική τροπολογία 3. Ξεκινάμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 73 τότε καταπίπτει και πάμε στην παράφα 10. Τροπολογία 75 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά επίσης απορρίπτεται. 77 υπέρ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας προφορίας. Πάλι ίδιο αριθμό ψήφων έχουμε, επομένω καταπίπτει αυτή η τροπολογία. Πάμε στην 76. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78. Νέα παράγραφος του κύριου Γκρέχ υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 80 της κυρίας Μακλάρκιν, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 79 του κυρίου Φόξ, υπέρ, κατά, επίσης απορρίπτεται. 81 Στάιλερ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 81. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18 υπέρ 17 κατά. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πολύ αργός. Ε, αν είχε ψηφίσει μπορεί να είχε επηρεάσει την, το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πιέσω κανένα. Μπορεί να είστε λίγο πιο έτσι γρήγοροι με το κουμπί σας. Ναι. Τέλο πάντων, περνάει με μία ψήφο υπέρ ε, επιπλέον. Επομένω η 82 καταπίπτει. Πάμε στην 83 του κ. Φόξ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 84 και 85. Ρούλερ και Στάιλερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 88. Στάιλερ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Α, απορρίπτεται. 80. Όχι, υιοθετείτε. Με δύο ψήφου υπέρ. Συγγνώμη κυρία Στάιλε, μπράβο, μπράβο. Οι 86 και 87 τότε καταπίπτουν. Σωστό, σωστά δεν τα λέω. Ναι, λέω ο Πάμε στα, στις αιτιολογικές σκέψεις. Έχουμε τις uh, τροπολογίες 1 και 2, που είναι οι ίδιες. Τις ψηφίζουμε υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά αυτές τις δύο τροπολογίες. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τρία της κυρίας Ρούλε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η τέσσερα καταπίπτει. Η πέντε του κύριου Γκρέχ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Η έξι και η επτά. Στάιλερ και Μακλάρκιν Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα αυτές τις δύο τροπολογίες 6 και 7. Πέρας. Απορρίπτονται. Άρα τώρα πάμε στην 8 και 10, Fox και Ρίλε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Πάλι ισοψηφία. Άρα καταπίπτουν και οι δύο. 9 Σμιτ. Ψηφίζουμε την 9. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 11 λοιπόν καταπίπτει. Πάμε στη 12 του κύριου Φόξ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 Στάιλερ. Υπέρ, όχι ηλεκτρονικά. Κατά. Γκρίνεται σαφώ. Η 13 λοιπόν καταπίπτει. 18 του εισηγητή. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 18. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 του κύριου Φόξ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 17. Αν δεν απατώμε. 17 της κ. Στάιλερ. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε εκτονικά. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Άρα, πάμε στο 16, Ρίλε. υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 19, η 19 λοιπόν καταπίπτει. Πάμε στην 20 του κύριου Φόξ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 22, Στάιλερ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. <coughs> Ένα μυστηριώδης πάλι δεν ψήφισε, αλλά τελείωσε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 18 υπέρ, 17 κατά. Θα μπορούσε να έχει αποφασίσει διαφορετικά αν είχε ψηφίσει αυτός ο μυστηριώδης τύπο. Εγκρίνεται πάντως 22 τη κυρία Στάιλερ. Πάμε στην τελική ψηφοφορία κατευθείαν λοιπόν. Α, πολύ αργά όπως και να είναι. Συγγνώμη. Καλή ισοψηφία είναι. Θέλει αυτός που αντικαθιστά τον εισηγητή να πει κάτι. Ο κ. Σταμπ. Όχι, όχι, τίποτα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν το σχέδιο γνωμοδότηση συνολικά. Έναρξη πληροφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Α, όλοι, αυτοί, όλοι ψήφισαν αυτή τη φορά. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 20 ψήφου υπέρ, 3 κατά και 13 εποχές. Ευχαριστώ κύριε Μάιε. Θα δούμε πώς θα συνεργαστούμε με την ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα, θα έχει ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να ενσωματωθούν οι τροπολογίες μας και να βρουν τη θέση τους και στην τελική ψηφοφορία. Θα προχωρήσουμε στη γνωμοδότηση του κ. Τριανταφυλλίδη για την ε, Ένωση της Καινοτομίας. Κυριάκο, επιθυμείτε να πείτε τίποτε. Σας ευχαριστώ. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω όλους τους και ηγητές για την συνεργασία τους, καθώς επίσης και τη γραμματεία για όλη την εργασία που κατέβαλαν. Όπως ε, γνωρίζετε, κάναμε μια πρώτη συνάντηση στην οποία συζητήσαμε τη γνωμοδότηση και προσπαθήσαμε να περιλάβουμε σε αυτήν όλες τις προφορικές προτάσεις που έγιναν εκείνη την ε, εποχή. Διατυπώσαμε σε αυτή τη βάση το πρώτο σχέδιο και μετά υποβλήθηκαν 49 τροπολογίες γραπτός. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους για την συμβολή τους που με βοήθησε πολύ. Το κείμενο εμπλουτίστηκε και μάλιστα τετραπλασιάστηκε σε μέγεθος. Η δική μου προσπάθεια πάντως ήταν πάντοτε να καταλήγω σε συμβιβαστικέ προτάσεις ώστε να καταστήσουμε ευκολότερη την ψήφιση της γνωμοδότησης. Εν τέλει 8 λοιπόν συμβιβαστικέ τροπολογίες. Η υπαριθμόν 1 δεν φέρει το όνομά μου αλλά κατά λάθο. Την υποστηρίζω απολύτως. Δυστυχώς δεν υποστηρίζω την 2 αλλά υποστηρίζω όλες τις υπόλοιπες συμβαστικές τροπολογίες και Πάλι ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία τους, για την παραγωγή νομίζω ενός εγγράφου, για τη σύνταξη ενός εγγράφου που ε, πραγματικά τιμά την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. ενώ το σημαντική γνωμοδότηση. Δείχνει την δέσμευση που έχουμε για το θέμα αυτό και που ε, είχε προσέλθει και η κυρία Γκιονκίνη να μας τα εξηγήσει. Πρώτα, τη συμβαστική τροπολογία, να ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2, ψήφι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 ως προσθήκη, υπέρ, κατά ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Προχωρούμε στην τροπολογία 26 υπέρ. Υπέρ. Υπέρ κατά, κατά εγκρίνεται άρα εκπίπτει 44. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται και αυτή. Προχωρούμε στην τροπολογία 36 του κυρίου Ρέπο. Εδώ έχει ζητηθεί κατά τμήματα. θα την ψηφίσουμε με τον τρόπο που, δείχνει που ε, ε, εδώ. Λοιπόν, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Α, συγγνώμη, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα τώρα, πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό όχι, υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Κατά. Εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε την 37, υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 9 υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή το τμήμα αυτό της ε, τροπολογικής ρέπο υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή. 45 κατά τμήματα πρώτο τμήμα της 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτό. 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 του κ. Γκρέκ Πάλι εδώ κατά τμήματα. Ψήφι υπέρ του τμήματος 1. Κατά. Εγκρίνεται. 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη με ψήφους 20 κατά και 15 υπέρ. Τροπολογία 4 υπέρ. 4 Αρχίζει η ψηφοφορία, ονομαστική τότε. Πέρας. Αυτή εγκρίθηκε. Παρόλο που δεν ψήφισε η κυρία Κόρχολα. 49. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43. Σουλή. Η... Μάλλον αρχίζει η ψηφοφορία ονομαστική. Πέρας. Απερίφθη. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, ονομαστική. Αρχίζει. That vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν 35 ψήφοι υπέρ, ούτε μία ψήφος κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, εξαιρετική εργασία πραγματικά και ελπίζω η αρμόδια ψηφιακή επιτροπή να αντιλάβει λάβει σοβαρά υπόψη της. Προχωρούμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. 11.30 έρχεται ο Επίτροπος. Έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο για την τελευταία αυτή ψηφοφορία. Ο κ. Άμπαντ είναι παρόν. Θέλετε να κάνετε μια εισαγωγή στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση λοιπόν για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών καθολικού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ όλες και όλους τους σκιώδης ηγητές, κολέγεται Κάμπος, Σμιτ, Κομφά και τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ για την συμβολή τους και την εργασία τους, καθώς επίσης ευχαριστώ και τη γραμματεία. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα κείμενο που είναι αρκετά συνενετικό και επιτρέπει να προχωρήσουμε στη συζήτηση σε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα λάβει υπόψη και την πολιτική σημασία που δίνουμε στην συνέχιση ύπαρξης α, καλής ποιότητας και σύγχρονων καθολικών υπηρεσιών. Η έκθεση του κ. Ντερόσα της Αρμόδιας Επιστοσίας Επιτροπή που έχει ήδη κατατεθεί και για 31 Μαρτίου προβλέπεται η προθεσμία κατάθεση τροπολόγιων. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να εγκριθεί η γνωμοδότησή μας, ώστε να ληφθεί υπόψη και από την αρμόδια ψηφιακή επιτροπή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας. Και νομίζω μάλιστα είναι η πρώτη σας γνωμοδότηση, που, η πρώτη γνωμοδότηση που κάνετε για λογαριασμό μας. Καλώς λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προχωρούμε λοιπόν στην τροπολογία 5 του κ. Τριανταφυλλίδη. Ψηφοφορία ονομαστική. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 6. Γκρέκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. επτά. επτά. Ανέμενα το σήμα σας κύριε Σφάμπ για να δω εάν θα κάνω τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας, πάλι το μυστηριώδες πρόσωπο δεν ψηφίσε, πάντως έχει απορριφθεί. Νομίζω ότι κάποιο δεν πατάει καλά το κουμπί, δεν το πατάει αρκετά δυνατά. Θα πρέπει να δείτε αν ανάβει το φωτάκι. Τέλο πάντων, τώρα αυτή απεριφθεί. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και προχωρούμε στην 13 του κ. Καμφάν. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 14, Γκρέκ. 14, δεν έχει πει υπέρ ο πρόεδρος. Τώρα λέει υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται σαφώς. Και τώρα 19 του κ. Γκρέκ. Αρχίζει η ψηφοφορία ονομαστική. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Και ακολουθεί η παριθμόν 26 ως προστίκη στην συμβαστική 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 27. Σμιτ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 28. Γκρέκ. Αρχίζει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθηκε αυτή. 29. Κρέκ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 33. Καφά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34. Καφά. Εδώ ζητείται ψηφοφορία κατά τμήματα. Άρα αρχίζει, ή μάλλον Ανοίγω την ψηφοφορία. Προς τα που θα πάτε, κύριε Σουάπ. Πρώτο λοιπόν μέρος, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απεριφθεί. Ψήφωσε επί του σχεδίου στο σύνολό του. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με ψήφους 34 υπέρ και 2 κατά και καμία αποχή. Ευχαριστούμε κύριε Άμπατ. Καλά λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους και όλους για την συνεργασία σας στις ψηφοφορίες. Προτείνω να διακόψουμε για λίγα λεπτά την ε, συνεδρίαση, αλλά παρακαλώ να είστε στις 11.30 εδώ για να μπορέσετε να θέσετε ερωτήσεις στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ταγιάννη, ο οποίος θα αναπτύξει το μελλοντικό πρόγραμμα των εργασιών του. Σας αναμένω στις 11.30. Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite you to uh, resume your places? We can resume the meeting. Ας επαναλάβουμε την συνεδρίαση, αφού σιγά-σιγά επιστρέφουν και οι συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά, με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Ταγιάννη, που φέρει την ευθύνη στο χαρτοφυλάκιό του για την ε, βιομηχανία και το επιχειρήν. Και βέβαια ε, έχει στα χέρια του πολλά σημαντικά θέματα της ενίας αγοράς που μας απασχολεί και πάντοτε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τον υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας διότι γνωρίζουμε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις εργασίες μας και αυτό ήταν και ο πρώην διαθρωμένος διάλογος μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω ότι έχει πια διαμορφωθεί καλή σχέση της Επιτροπής μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην χρειαζόμαστε τον διαθρωμένο διάλογο, να είμαστε σε διαρκή διάλογο πλέον. Ορισμένες φορές βεβαίως είμαστε επικριτικοί, αλλά πάντοτε με επικοδομητικό πνεύμα. Συζητήσαμε ήδη σήμερα ορισμένα θέματα για τα γεωργικά μηχανήματα, τους γεωργικούς ελκυστήρες και το απόγευμα έχουμε ακρόαση για τις μοτοσυκλέτες και τα άλλα σχετικά δίκυκλα. Θα μας αναπτύξετε τα σχετικά με το πρόγραμμά σας, μετά οι συνάδελφοί μου θα μπορέσουν να σας θέσουν ερωτήσεις και εσείς βεβαίως θα έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Σας δίνω το λόγο λοιπόν, αφού σας καλωσορίσω για μια φορά ακόμη. Ευχαριστώ, Μάικλ. Κάθε φορά που έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, έρχομαι με μεγάλη χαρά. Το Κοινοβούλιο μένει στην καρδιά μου μετά από τόσα χρόνια που πέρασα σε αυτά τα έδρανα. Πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή η σχέση είναι πολύ σημαντική. Όπως θα ξέρετε, φέτος προώθησα μια σειρά από πρωτοβουλίε σημαντικές για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ τη βιομηχανία, Όπως ξέρετε, ο στόχος μου ο βασικός είναι να θέσω στο κέντρο των πολιτικών μας πρωτοβουλειών την πραγματική οικονομία. Και πραγματική οικονομία σημαίνει πάνω απ' όλο ανάπτυξη της αγοράς, της εσωτερικής αγοράς. Επομένω, θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιε δράσει μέχρι το τέλο τη νομοθετική θητεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί θεωρώ ότι μετά την κρίση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερβούμε τις δυσκολίες, να ανακαλύψουμε ξανά την πραγματική οικονομία, γιατί αυτό είναι το πραγματικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει. Με μεγάλη ικανοποίηση πρέπει να πω οι τέσσερι στρατηγικέ πρωτοβουλίε που είναι κάτω από την ευθύνη μου και που προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν για το 2010 και 2011. Από αυτέ, δύο έχουν ήδη υιοθετηθεί το 2010 και αφορούν την Ένωση για την Καινοτομία, που είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που με μεγάλη χαρά ε, προώθησα μαζί με την συνάδελφό μου, την ε, Επίτροπο Γιώργαν Κουίν, και τη νέα ε, βιομηχανική πολιτική. Αυτές είναι οι δύο βασικές πρωτοβουλίες. Οι άλλες δύο αφορούν την τυποποίηση που θα υιοθετηθεί μεταξύ Απριλίου και Μαΐου του 2011 και η τέταρτη είναι η στρατηγική για, την, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2011. Τώρα, εργαζόμαστε επί μιας άλλης στρατηγικής ε, πρωτοβουλίας ε, που είναι το Single Market Act που είναι αρμοδιότητας του κυρίου Μπαρνιέ ε, ενεπλάκην όμως εκ του σύνεγγυς, γιατί είναι υπεύθυνο για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Και μεταξύ των ε, πρωτοβουλειών που θα υιοθετήσει τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, εγώ προωθώ δύο στοιχεία για, που μου φαίνονται σημαντικά για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς. Την πρόσβαση στις πιστώσεις από τη μία και την γενική ασφάλεια των προϊόντων, από την άλλη, που είναι στοιχεία που αναφέρονται και στην πρόσφατη αναθεώρηση που έγινε, που είναι ένα άλλο σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση και πρόθεση όλων των προϋποθέσεων, τόσο ώστε οι, μικρές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποφεληθούν πλήρως από την εσωτερική μας αγορά. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση, από τις 11 προβλεπόμενες πρωτοβουλίες, οι τρεις έχουν ήδη υιοθετηθεί. Οι τέσσερις προβλέπεται να υιοθετηθούν μέσα στο 2011 και οι υπόλοιπε ε, τέσσερις θα υιοθετηθούν μέσα στο 2012. Συνολικά, η συνεισφορά μου πιστεύω ότι θα είναι αποφασιστική για το πρόγραμμα απλούστευσης που προωθεί συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος σήμερα είναι να κάνω μια επισκόπηση μαζί σας ε, και να σας παρουσιάσω τις πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί για το υπόλοιπο του 2011 και για τον επόμενο χρόνο, το 2012. Θα σας μιλήσω για την εποπτεία της εσωτερικής αγοράς, την τυποποίηση, για πρωτοβουλίες για τα αυτοκίνητα και θα σταθώ πιο συγκεκριμένα στο θέμα της έκδοσης πινακίδων. Επίσης, θα μιλήσω και για πιλωτικά σχέδια καινοτόμα στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων και θα σας δώσω και κάποιες πληροφορίες που αφορούν κάποιες πρωτοβουλίες κλειδιά επί των οποίων εργαζόμαστε, που είναι τα κλώστα φωτοβουλικά και η οδηγία για τα παιχνίδια. Και η εφαρμογή στα κράτη-μέλη της οδηγίας αυτής για τα, παιχνίδια. Θέμα αρκετά ευαίσθητο και θα σας δώσω κάποια νέα, κάποιες ειδήσει που δεν είναι πολύ θετικά. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς. Αυτό το θέμα προφανώς είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, είναι βασικό για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η θέση σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2010 του κανονισμού 765 του 2008 σε ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς ε, συνεισέφερε σημαντικά για να προωθήσουμε την πολιτική μας σε αυτόν τον τομέα και να αφήσουμε ένα σημαντικό αποτύπωμα. Με τη θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού, η εποπτεία της αγοράς εντοπίστηκε ως προτεραιότητα που θα πρέπει να την προωθήσουμε σε επίπεδο ένωσης, όχι μόνο με την πρόσφατη μου ανακοίνωση για τη νέα ε, βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης, αλλά και με την ανακοίνωση προς μία πράξη, ένα νομοθέτημα δηλαδή, για μία ενιαία αγορά. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς, ε, Πρόεδρε και η Επιτροπή σας, υποστηρίζετε έντονα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την προσπάθεια που σκοπό έχει να βελτιώσει και να ενισχύσει το σύστημα ελέγχων για τα εισαγόμενα προϊόντα ή για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση της ε, κυρίας Σαντεμόζα που υιοθετήθηκε αυτό το μήνα και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ακολούθησε είναι η πιο σαφής μαρτυρία. Προσωπικά είμαι πεπισμένος, μια και πρότεινα ή μάλλον όπως προτείνετε εσείς σε αυτή την έκθεση Σαλντεμόζε, ότι είναι σημαντικό να διαθέτουμε ένα ενιαίο σύστημα παρακολούθησης που να αφορά όλα τα προϊόντα που προορίζονται σε καταναλωτές ή σε επαγγελματίε, είτε είναι αρμονισμένα είτε όχι. Ένα ενιαίο σύστημα θα έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα προς τους καταναλωτές, που έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε, προς τις εθνικές αρχές που πρέπει να έχουν τα απαραίτητα μέτρα για να εποπτεύσουν αποφασιστικά την αγορά, αλλά θα πρέπει επίση να υιοθετήσουν και οικονομίες κλίμακας και προς τους οικονομικούς φορείς που θα έχουν την εγγύηση ότι θα υφίστανται ένα θεμητό ανταγωνισμό. Για, σε ό,τι με αφορά, είχα την ευκαιρία να σας ενημερώσω τον περασμένο Νοέμβριο ε, και στο, την επιστολή προς τον ε, πρόεδρο Χάρμπουρ έδειξα τη σημασία που έχει η ενίσχυση αυτού του πυλώνα στην νομοθετική διαδικασία. Θα σε ενημερώνω για όλες τις δραστηριότητε ε, που έχουν ήδη ξεκινήσει και για τις μελλοντικέ. Καταρχά, είμαι πεπισμένο ότι είναι απαραίτητο να καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια για να καταστήσουμε ισοδύναμα και συγκρίσιμα τα μέτρα των εθνικών αρχών καθώ και τα μέτρα ελέγχου που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. το στόχο αυτό δεν μπορούμε να τον επιτύχουμε με σποραδικέ δράσει και με ad hoc δράσει. Θα πρέπει να έχουμε του απαραίτητου πόρου και μια προσέγγιση συνεπή. Πέρα από την έγκριση με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη νέα πολιτική που είναι δύσκολο έργο, περίπλοκο και θα απαιτήσει ε, προσπάθεια συντονισμού από πλευρά κομισιών για να αποφύγουμε διαφορέ κενά και παραλήψεις, θα ήθελα να σα αναφέρω τρει δράσει ε, που θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα. Καταρχά, θα πρέπει να έχουμε ένα γενικό πολιετές πρόγραμμα, όπου πέρα από τις δραστηριότητες οργάνωσης ε, και εποπτείας της αγοράς θα αναφέρουμε με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να δούμε τις ανάγκες, τα μέσα και τους τρόπους, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την εποπτεία τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτά τα βασικά στοιχεία του προγράμματος τα επεξεργαζόμαστε ήδη σε αυτή τη φάση. Η Κομισιόν θα πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσει συγκεκριμένες αποφάσεις μέχρι το τέλος ε, του 2012. Η δεύτερη δράση προτεραιότητας θα πρέπει να προβλέψουμε την αναθεώρηση του συνολικού νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς. Όντω, ε, εξετάσουμε τη δυνατότητα να επανεξετάσουμε μέχρι το τέλο του 2011 την οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων, ούτω ώστε να έχουμε ένα κείμενο και να έχουμε εκεί όλα τα στοιχεία εποπτεία αγορά ε, που υπάρχουν σε εκείνο τον κανονισμό και στον κανονισμό 765 του 2008. Έτσι θα έχουμε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, ένα ενιαίο σύστημα ε, που να συνάδει με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με τα ψηφίσματα, με το ψήφισμα μάλλον που υιοθετήθηκε αυτό το μήνα. Η τρίτη δράση. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου μέσω κάποιων οριζόντιων πράξεων. Φερρυπίν. Μέσω μιας αποτελεσματικής συνεργασίας μαζί και μέσω των τελωνίων, θέτοντας σε ισχύ μια ισχύ, κοινή μεθοδολογία για τον καθορισμό των κινδύνων, να δούμε τα προγράμματα ε, τα εθνικά εποπτείας, αλλά και μέσω μιας ε, συνεπούς δράσεως και μιας κατάλληλης διοικητικής συνεργασίας. Αυτές οι δράσεις ε, θα μεταφραστούν στην πράξη στους διάφορους βιομηχανικούς τομείς που καλύπτει ο καονισμός 765. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το 75% των προϊόντων των βιομηχανικών, τα παιχνίδια, τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, οι ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Όλα αυτά θα τα καλύψουμε. Και πάμε τώρα στο σήμα CE. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για εποπτεία τη αγορά χωρίς να μιλήσουμε για το σήμα CE. Είναι ουσιώδες για τη σωστή λειτουργία τη εσωτερική αγορά και για την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, γιατί στέλνει ένα μήνυμα αποτελεσματικότητα του κανονιστικού μας συστήματο ό,τι αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Ε, κατόπιν αιτήματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κομισιόν ε, δεσμεύτηκε να προωθήσει μια εκστρατεία ενημέρωση για το σήμα που θα αφορά του ε, οικονομικού φορεί ε, γενικά και κυρίω εκείνου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και να καλύψουμε και του καταναλωτέ. Η Κομισιόν ξεκίνησε αυτή την εκστρατεία στι αρχέ του 2010 και είναι πολύ ικανοποιημένη και από την εξέλιξη και από τα αποτελέσματα αυτή τη εκστρατεία. Όλα τα στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν ότι πάει καλά αυτή η προσπάθεια, είναι θετικά. Μετά από την υιοθέτηση του νέου κανονιστικού πλαισίου για την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εμπορευμάτων το 2008, το Κοινοβούλιο μου ζήτησε κατ' επανάληψη να εξετάσω τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα ευρωπαϊκό σήμα για την προστασία των καταναλωτών. Προς το παρόν, όπως είπα και στην τελευταία συζήτηση που κάναμε εδώ στο Κοινοβούλιο, που τέθηκε αυτό το θέμα, είμαι πεπισμένο ότι η αξιοπιστία του σήματο και η ασφάλεια των προϊόντων είναι θεμελιώδου σημασία για μια αποτελεσματική εποπτεία τη αγορά ε, που είναι σημαντική σε μια πρώτη φάση και επομένω θα πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε πρώτη φάση για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Παρ' όλα αυτά, είμαι στην διάθεσή σας για να επανεξετάσουμε το σύστημα ε, σήματος στα πλαίσια της έκθεσης της Επιτροπής που θα σας παρουσιάσει η Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2013 για την ενεργοποίηση του κανονισμού 765 του 2008. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευθυγράμμιση των 10 οδηγιών του νέου νομοθετικού πλαισίου με σκοπό να εφαρμόσουμε το πακέτο προϊόντων πολύ γρήγορα, η Κομισιόν ετοιμάζει μια σειρά από προτάσεις που θα υιοθετηθούν μέχρι το καλοκαίρι που σκοπό έχουν να ευθυγραμμίσουμε 10 οδηγίες που αφορούν τα προϊόντα με την απόφαση 768 του 2008. Πάμε στην τυποποίηση. Έχουμε συζητήσει ξανά αυτό το θέμα τον Ιούνιο του 2010 όταν έγινε αυτή η ακρόαση που οργανώθηκε από τον πρόεδρο Χάρμπορ και από την Επιτροπή. Ε, τότε σας είπα ότι η Κομισιόν ετοίμαζε, ένα σχέδιο να αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Τυποποίησης και σας επιβεβαιώνω τώρα ότι λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης καθώς και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου του 2010 για το μέλλον της τυποποίησης. Το ψήφισμα που μας έστειλε ένα μήνυμα πολύ ξεκάθαρο. Αναθεώρηση. Αλλά όχι επανάσταση. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι η προτινόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να βασιστεί στα βασικά, στα ισχυρά σημεία του σημερινού συστήματος και να αποφύγει ρηξικέλευθες αλλαγές. Καμία επανάσταση λοιπόν. Τέλο πάντων, θα πρέπει παρόλα αυτά να καλύψουμε τα κενά, γιατί υπάρχουν κενά στο σύστημα. Όπω υπογραμμίσατε, διαδικασίες τυποποίησης είναι πολύ αργές και πολύ περίπλοκες. Πέρα από την ε, βελτιωμένη συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, θα πρέπει να εμπλέξουμε και του καταναλωτέ που ενδιαφέρονται για τη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν μεταξύ Απριλίου και Μαΐου θα υιοθετήσει μια στρατηγική ανακοίνωση για την τυποποίηση, καθώ και μια νομοθετική πρόταση. Ο βασικός στόχος των δύο αυτών κειμένων είναι να βελτιώσουμε την λειτουργία τη εσωτερική αγορά να επιταχύνουμε και να εκμοντερνήσουμε τι διαδικασίε τυποποίηση για να υπάρχει διαλειτουργικότητα και για να προωθήσουμε την καινοτομία στην παγκόσμια αγορά που εξελίσσεται εντάχει. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των αυτοκινήτων, έχουν γίνει πάρα πολλά και γίνονται ακόμα πολλά. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε δύο στοιχεία, την έκδοση πινακίδων και την νομοθεσία που έχουμε ήδη δρομολογήσει. Ας ξεκινήσουμε από την καταχώρηση των αυτοκινήτων. Οι πολίτε και οι επιχειρήσει εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίε ό,τι αφορά τη μεταφορά των οδηγίων, τα οποία είχαν πινακίδε σε ένα άλλο κράτο μέλο και θέλουν να τα μεταφέρουν σε ένα άλλο κράτο μέλο. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη επιβάλλουν στα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν μονίμως ε, στην επικράτειά τους να λαμβάνουν ε, πινακίδες από τις εθνικές αρχές με βάση εθνικούς κανόνες. Αυτό ε, σημαίνει ότι όταν ένας πολίτης ή μια επιχείρηση θέλουν να πάνε σε άλλο κράτος μέλος, το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαγραφεί από το Μητρό των κρατών μελών και να ξανακαταχωρηθεί στο σχετικό μητρό του νέου κράτος μέλους. Η διαδικασία διαγραφής χαρακτηρίζεται συχνά από τρομερές καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια. Ε, ζητούμε τεχνικές πληροφορίες ε, επιπλέον. Καμιά φορά το άτομο δεν μπορεί να απαντήσει και επομένως ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν δεν θέλετε να χάσετε χρόνο, κανονικά πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα ειδικό για να σας ρυθμίσει αυτό το θέμα. Αυτό επιφέρει όμως κόστος για τους πολίτες. Για να καλύψουμε αυτό το πρόβλημα στην εσωτερική αγορά μέχρι το τέλος του 2011. Η Κομισιόν θα υιοθετήσει νέες πρωτοβουλίες που θα απλουστεύσουν τους τρόπους και τις προϋποθέσεις ε, καταχώρησης των αυτοκινήτων που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε ένα άλλο κρατός μέλος. Αυτό το κείμενο είναι μία από τις ε, δράσεις που αναφέρονται στην έκθεση του 2010 για την ηθαγένεια και ε, εντάσσει την πράξη για την ενιαία αγορά του 2010. Στις 3 Μαρτίου 2011 η Κομισιόν ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση που τελειώνει στις 26 Μαΐου ε, για να δούμε ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την καταχώρηση των αυτοκινήτων. Η διαβούλευση, αυτή θα δείξει ποιες είναι οι απόψεις των ε, πολιτών και των ενδιαφερομένων και σκοπό έχει βεβαίως να φύγουν τα εμπόδια ε, στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, των εμπορευμάτων, των αυτοκινήτων τώρα. Τώρα, για την νομοθεσία για τα αυτοκίνητα. Ας ξεκινήσουμε από την απλούστευση ε, της νομοθεσίας ό,τι αφορά την ε, τυποποίηση των αυτοκίνητων. Τα τελευταία χρόνια το νομοθετικό πλαίσιο για την τυποποίηση υπέστη μια έντονη προσπάθεια απλούστευσης. Ε, και το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ε, ο σημαντικό, η σημαντική μείωση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων. Έχουμε μία βασική ε, οδηγία, την οδηγία πλαίσιο 2007-46 και από 7 ε, ξεχωριστούς κανονισμούς. Το κανονιστικό πλαίσιο για τα οχήματα κατηγορίας L και για τους ελκυστήρες, δηλαδή μοτοσυκλέτες και ελκυστήρες, ε, θα ακολουθήσει το ίδιο μοντέλο. Και η Επιτροπή το 2010-2011 υιοθέτησε τέσσερις προτάσεις στα πλαίσια της συναπόφασης που αυτή τη στιγμή τη συζητάμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Όλο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό, μια σημαντική προσπάθεια έτσι, απλούστευσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως σας είχα ανακοινώσει στην ε, στρατηγική για τα καθαρά οχήματα και οικολογικά οχήματα τον Απρίλιο του 2010, θα πρέπει να έχουμε μέτρα γενικού χαρακτήρα, ώστε να εφαρμόσουμε κοινά κοινού κανόνε στα ηλεκτρικά οχήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2009 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπόκεινται σε μια ευρωπαϊκή τυποποίηση, όπω και τα άλλα ε, συμβατικά οχήματα. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί σε επίπεδο της UNECE, που είναι η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ, προκειμένου να καθορίσει τους τεχνικούς κανόνες για τα ηλεκτρικά οχήματα και μπορώ να σας πω ότι έχουν ε, σημειωθεί μέχρι τώρα σημαντικά βήματα, σημαντική πρόοδος. Ε, έχουμε όλα τα στοιχεία ε, που μας χρειάζονται για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ενίας αγοράς για τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και με αυτή την προσέγγιση θα εξασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσει Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι οι ίδιες με εκείνες που έχουμε συμφωνήσει σε διεθνές επίπεδο. Πάμε τώρα στις νομοθετικές προτάσεις που ετοιμάζουμε στον τομέα του αυτοκινήτου για φέτος. Καταρχάς, μιλάμε για τον, για τον ήχο που εκπέμπουν τα οχήματα με κινητήρα, ε, κανόνες για τις εκπομπές, καλύτερη υποπτία της αγοράς και διάφορα μέτρα σε περίπτωση που υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ οδηγεί κανείς αυτά οχήματα. Τώρα πάμε στα κλωστοϊφαντουργικά. Θα του αρέσει αυτό του Προέδρου. κάνει κάποια γλωσσικά σχόλια που αφορούν τα Ιταλικά ο κ. Σταγιάννη. Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την αντικειτοθεσία των κλωστοϊφαντουργικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ακόμα μια φορά την Επιτροπή σας και κυρίως τον κύριο Μάντες για την έντονη προσπάθεια που έκανε για το θέμα, για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια τη πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Επαναλαμβάνω την υποστήριξη της Επιτροπής προς τις ε, τροπολογίες του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων και για την, το σήμα προέλευσης και τις ενδείξεις που αφορούν ε, στοιχεία ζωικής προέλευσης. Και εγώ προσωπικά και η Κομισιόν θέλουμε να συνεισφέρουμε στην, ε, στις διαπραγματεύσεις τώρα που φτάνουμε σε μια κρίσιμη φάση της δεύτερης ανάγνωσης. Θα πρέπει να αντικοπήσουμε τις συζητήσεις για πολιτικά ευαίσθητα θέματα και κυρίως αυτό που αφορά το σήμα προέλευσης, ούτως ώστε, η καταγωγής, ούτως ώστε να φτάσουμε σε συμβιβασμό μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ή δυνατό στα πλαίσια της δεύτερης ανάγνωσης. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ πιο περίπλοκο θέμα που είναι τα παιχνίδια. Δεν είναι κάτι που πιστεύω μόνο εγώ προσωπικά, αλλά είναι μια δέσμευση που έχει λάβει η δυνατο στα πλαισια τη δεύτερη ανάγνωση. και παμε τωρα σε ενα πολυ πιο περιπλοκο θεμα που ειναι τα παιχνιδια Επιτροπή. Ε, δηλαδή ότι το θέμα των ε, συμφερόντων των καταναλωτών των πιο ευπαθών, που είναι τα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό για μας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η οδηγία για τα παιχνίδια που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2009, που ενισχύει τους κανόνες ασφάλειας σε ό,τι αφορά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Ήδη συζητήσαμε πολύ εκτεταμένα αυτό το θέμα, ε, όταν ε, παρουσιάστηκε σχετική ερώτηση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Θα ήθελα τώρα, επ' ευκαιρία της σημερινής ε, παρουσίας μου εδώ, να σας, κάνω, να σας δώσω κάποια νέα στοιχεία. Όπως έχω πει πολλές φορές, ε, θέλουμε μέσω της επιτροπολογίας να εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση της ε, νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τι επιστημονικέ και τεχνολογικέ εξελίξει, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά την, το κατάλληλο επίπεδο προστασία. Αυτή η δουλειά έχει ξεκινήσει ήδη για τι ουσίε που μα ανησυχούν πολύ όπως το κάδμιο και ο μόλιδο, Η ομάδα των ε, εμπειρογνωμόνων θα συνεδριάσει εκ νέου 4 και 5 Απριλίου του 2011 για να συζητήσει τα, τις χημικές ενώσεις, χημικέ χημικές ουσίες. Και με βάση την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων η Κομισιόν θα προτείνει μέτρα επιτροπολογίας για το κάδμιο, τον, το μόλιδο μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 και άλλα μέτρα για την τροποποίηση της των τοξικών ουσιών, καρκινογενών ουσιών και μεταλλαξιογόνων ουσιών μέχρι τις αρχές του 2012. Για να όσο αυστηρή και να είναι πάντως η νομοθεσία, εάν δεν ε, γίνει σεβαστή, δεν αρκεί. Είχαμε 10 συνεδριάσεις ε, σε ομάδες εργασίας για τα παιχνίδια με τις κινέζικες αρχές. Και έχουμε και μια ομάδα εργασία για τα παιχνίδια με αρχέ από τι ΗΠΑ, ούτω ώστε να ενημερώσουμε και τη χώρα αυτή για τα νέα μέτρα. Τέλος, ένα νέο που για μένα δεν είναι θετικό, υπάρχει μια διαδικασία επιπαραβάση. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να το παίζει τιμωρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μου αρέσουν αυτά τα νέα αλλά ό,τι και να κάναμε ε, ήταν μάτιν. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε μια διαδικασία επί παραβάση απέναντι σε 17 χώρες. Γιατί δεν ε... εφάρμοσαν σωστά την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πιλωτικά σχέδια, τα καινοτόμα για τις δημόσιες προμήθειες, είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον πρόεδρό σας, τον κύριο Χάρμπορ. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της ομιλίας μας. Πριν τελειώσω όμως, θα ήθελα να προσθέσω τι ακριβώς έχουμε κάνει. Για να υποστηρίξουμε τις ε, δημόσιες υπηρεσίες ε, στον τομέα των ε, αγαθών και υπηρεσιών και τόμο χαρακτήρα. Νομίζω εδώ τα νέα είναι θετικά. Ένα δωράκι για τον πρόεδρο. Σας υπενθυμίζω ότι στο πλαίσιο της Ένωση για την Καινοτομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να δώσει οικονομική υποστήριξη και προσανατολισμό στι ευρωπαϊκέ αρχές που θέλουν να προωθήσουν την καινοτομία. Συνεστάσει στα κράτη-μέλη να κρατήσουν ένα τμήμα από τα κονδύλια τους για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καινοτόμου χαρακτήρα. Στι 4 Φεβρουαρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα καθεστώ έρευνα και καινοτομία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Γι' αυτό ε, οι υπηρεσίε μου μαζί με την ε, Γενική Διευθύνση και το RTD τη Κομισιόν ξεκίνησε μία μελέτη σκοπιμότητα για, για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ένα ε, ευρωπαϊκό καθεστώ υποστήριξη των ε, δημοσίων προμηθειών υπέρ τη καινοτομία. Αυτό τι σημαίνει. Από τη μία, προϊόντα τα οποία ε, μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά, που δεν χρειάζονται κατά, ανάγκη έρευνα και ανάπτυξη. Κατά την άλλη, ε, υπηρεσίες που δεν υπάρχουν, που απαιτούν έρευνα και ανάπτυξη μέσω α, ε, προεμπορικού χαρακτήρα. Στην πρώτη φάση αυτής της μελέτης, ορισμένοι από συμμετείχαν. Αυτό το σύστημα ε, συνδέει ε, τις δημόσιες προμήθειες ε, προϊόντων που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά ε, με διαγωνισμούς προεμπορικού χαρακτήρα. Θα υπάρξει υποστήριξη από την Ευρώπη για, τις, για τους διαγωνισμούς, σε πάση υπέρ της καινοτομίας. Προβλέπουμε 15 ε, εκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα το ανακοινώσουμε στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής διάσκεψης που θα γίνει ε, στο τέλος του Ιουνίου στο Τωρίνο. Θα δούμε τώρα αν χρειάζονται νομοθετικές προσαρμογές, ούτως ώστε να υπάρξει ε, ένα τέτοιο καθεστώς ευρωπαϊκό σε μεγάλη κλίμακα μετά το 2013. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία των κοινών διαγωνισμών που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την καταπολέμηση της, του, του κατακαιρματισμού της ζήτησης και για την υποστήριξη της εσωτερικής αγοράς, που δεν, αγορά η οποία δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη στην Ευρώπη, λόγω του ότι ε, το πλαίσιο, το κανονιστικό δεν είναι σωστό. Τα αποτελέσματα ε, θα σας τα ανακοινώσουμε τον Αύριο του 2011. Θα είναι ένα χριστουγεννιάτικο θόρο για τον Πρόεδρο και ελπίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας επιτρέψουν αυτά τα αποτελέσματα να υιοθετήσουμε ένα πραγματικό καθεστώς ευρωπαϊκό ε, υποστήριξης των ε, διαγωνισμών καινοτομία. Και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουμε τις προσπάθειες που κάνουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Μην ξεχνάτε τη δουλειά που έκανε ο Μπαγνιέ και το Green Paper, την πράσινη βίβλο δηλαδή, για τις, τους διαγωνισμούς αυτούς. Ξέρω ότι μακρηγόρησα, αλλά προσπάθησα να σας δώσω όλες τις πληροφορίες που έχω για τα θέματα της αρμοδιότητάς μου που ενδιαφέρουν την Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για την υπομονή σας. Yeah. Well, I think, uh... νομίζω, νομίζω, αντιπρόεδρε, Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό, διότι μια ολόκληρη σειρά πρωτοβουλειών αναπτύσσονται και πολλές ανταποκρίνονται στα αιτήματα που είχαμε διατυπώσει εμείς και έτσι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ως έκθεση. Πολλή δουλειά έχουμε να κάνουμε και χαίρεται η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή να αναλάβει αυτό το έργο. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση και με τις παρεμβάσεις. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, σε ομάδε τριών θα γίνονται οι παρεμβάσει να έχουμε καλύτερα διαμορφωμένο διάλογο με αυτόν τον τρόπο. Αυτή τη στιγμή έχω, για να δούμε ποιοι θα ήθελαν να παρεμβάσουν. Θα σα πω ποιοι είναι στου αγορητέ. Και μετά μπορούν να προσθεθούν ονόματα για να κατανεμηθεί ο χρόνο. Professor Κύριο Σαμπάτ. Άλλη. Η Και η κυρία Ράπτη. Άλλη, παρακαλώ. Right, okay. Πολύ καλά. Λοιπόν, ένα λεπτό περίπου καθένας ε, ώστε να έχουμε μια σύντομη έτσι, παρέμβαση από τα ερωτήσεων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι σε μισή ώρα θα μπορούν να παρέμβουν. Συμφωνείτε. Ε, δύο λεπτά κατά το μέγιστο, εντάξει, ω όριο. Και ο κύριος Μπούσουτη λυπούμε και, και εσείς κύριε. Πόσους έχουμε. Εντεκά uh, συνάδελφοι. Αν είσαστε σύντομοι, ένα λεπτό καθένα, τότε θα ήταν τέλειο. Και αυτό θα σα αναφέρω σε σχέση με το χρονόμετρο όταν θα έχετε φτάσει στο όριό σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι πάντα χαρά να έχουμε ανταλλαγή απόψεων μαζί σα. Είμαι ως αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, και αυτά πήγαν καλά. Σας ευχαριστούμε. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως πρώτον. Το είδαμε στην κρίση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι η ραχοκοκαλιά ακριβώς της οικονομίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό όλες οι προσπάθειες από πλευρά σας το γραφειοκρατικό βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μειωθεί, αλλά και να είναι ανταγωνιστικές στην αγορά. Όλες οι πρωτοβουλίες σα ε, είναι καλοδεχούμενες σε μεγάλο βαθμό και η ομάδα του έλθανε πάντα στο πλευρό σας όταν συνεχίζετε αυτό το έργο. Αναμένουμε δεύτερον με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση για την ευρωπαϊκή τυποποίηση και με θετικό τρόπο σημειώσαμε ότι καταφέραμε σε σχέση με τις συσκευές να ενταχθούν ε, και αυτές και να έχουμε και πρότυπα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετηθούν από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε σε αυτό το εγχείρημα, διότι θα μπορούσαν να αποκομίσουν μεγάλα ωφέλη οι καταναλωτές. Τρίτον, η οδηγία για τα παιχνίδια. Το βρίσκω πολύ θετικό ότι θα ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση έναντι των κρατών μελών όταν δεν τηρούν τι διαδικασίε στα κράτη-μέλη. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα ότι οι σημερινέ προδιαγραφέ είναι υψηλότερε από αυτέ που έχουν αποφασιστεί και γι' αυτό με τη διαδικασία επιτροπολογία θετικό είναι να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Θα είναι δύσκολο όμω για αυτέ τι χώρε να μειώσουν, να χαμηλώσουν το επίπεδο προστασία από πλευρά των προδιαγραφών του και μετά να το ανυψώσουν. Θα είναι εύκολο ίσω με τη διαδικασία επιτροπολογία, σα να αποφύγουμε κάτι τέτοιο και να διευθετήσουμε τα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Σουβάπ. Ο καθηγητής Κορέιντερ Κάμπο έχει τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Επίτροπε που ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στην κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Πολύ σύντομα κάποια σημεία σε σχέση με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την γενική ασφάλεια των προϊόντων. Σε μια επίσκεψη που έκανε η Επιτροπή ΙΝΚΟ και σε επαφές με τους Ούγγρους βουλευτές ε, που ήταν τα πιο σημαντικά σημεία αυτά παράπονα για την ποιότητα ακριβώς των προϊόντων. Εμείς, εσείς αναφέρατε ότι θα υπάρξουν οριζόντιες εγκάρσιες δράσεις ε, ώστε να επιτραπεί να είμαστε πιο αποτελεσματικοί Υπάρχει μια τάση, δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό, υπάρχουν κάποιες φήμες που κυκλοφορούν ότι κάποιες τρίτες χώρες αποκτούν ή προχωρούν στην ε, διαχείριση κάποιων μεγάλων λιμένων στην Ευρώπη, κυρίως ε, στην ε, νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ερωτώ, διαρωτώ με αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια πρόσθετα ίσως προβλήματα για τις εγγυήσεις της ασφάλειας των προϊόντων στα σύνορα της Ένωσης. Δεύτερη ερώτηση, για τα οχήματα, κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα, η δεύτερη ερώτηση. Κάνατε λόγο για μία τέτοια καταχώρηση όσον αφορά τις προδιαγραφές. Υπάρχουν κάποια σχέδια για ένα για τον, την εξομάλυνση της ε, διαδικασίας ε, της φόρτισης ε, μπαταριών των συσσωρευτών βραχυπρόθεσμα γιατί θα πρέπει με βάση αυτούς τους μηχανισμούς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια ερώτηση ακόμα μιλήσατε για μέτρα όχι μόνο για χρηματοοικονομικούς πόρους, αλλά επίσης και για την ανάγκη νομοθετικών πλαισίων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για το πρόγραμμα ε, Εύρικα, Eureka, σε σχέση με τις χώρες ε, που εμπλέκονται και για τρίτες χώρες επίσης, πέρα από τους, ε, τα 27 κράτη-μέλη. Ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε, δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημαντική πείρα όσον αφορά την καινοτομία και όσον αφορά και τη διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρω ότι υπήρχαν πολύ στενές σχέσεις σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να ξέρω, υπάρχει κάποια δυνατότητα από το Εύρικα να γίνει κάτι. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Um... Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπουσόη, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστούμε για τις προσπάθειες ε, να υπάρξει ε, ένα κοινό πλαίσιο για την διεύρυνση με την ενιαία εσωτερική αγορά αυτών των διατάξεων. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία φυσικά που υιοθετείται ε, θα είναι σημαντική για την ενιαία εσωτερική αγορά. Και έτσι σίγουρα θα προσθέσει πρόσθετη αξία. Παρ' όλα αυτά παραμένουν κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν στενότερης ε, εκ του σύνεγγης προσοχής ε, για τα προτερήματα που θα απορρεύσουν για τις ε, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πραγματικά στην δική μου έκθεση για την ενιαία εσωτερική αγορά για τις επιχειρήσεις, μία από τις προκλήσεις όταν έχουμε το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζουμε, είναι μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απολάβουν όλων των προτεραιμάτων της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Το γεγονός... Αναθεώρηση του Small Business, του ε, Small Business Act είναι πολύ σημαντικό για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε έτσι πολλά μέσα χρηματοδότησης, ε, όπως και αυτά που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Παρ' όλα αυτά, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν όλες αυτές τις ευκαιρίες και πολύ πιθανόν η Κομισιόν θα έπρεπε να κάνει κάποιες προσπάθειες ούτως ώστε να ευαισθητοποιήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέρα από το, σχέδιο για να βελτιώσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κεφάλια στις κεφαλαγορές, θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για αυτό το σχέδιο δράσης για την πρόσβαση στις χρηματαγορές ε, και ποιε είναι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά. Αυτό, μαζί με τη μείωση των διοικητικών βαρών, ε, είναι πολύ σημαντικά για να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες μας επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο καινοτόμε. Ευχαριστώ. Καλά, θα παρακαλέσω τον Επίτροπο να απαντήσει πρώτα σε, αυτής, σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και μετά θα προχωρήσουμε αναλόγως με τον χρόνο που μας μένει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω πάρα αυτά. Ε, θα σας εξηγήσω τι κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουσό για τα θαυμάσια ιταλικά σας. Με ευχάρισε πάρα πολύ που σας άκουσα μιλάτε ιταλικά. Εγώ δυσκολεύομαι πιο πολύ να μιλήσω τη δική σας μετρική γλώσσα, είναι πιο περίπλοκη. Τέλος πάντων. Εμεί δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί όπω είπε και ο κ. Σφαπ, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα τη οικονομία μα. Αν θέλουμε λοιπόν, όπω είπα και στην αρχή, να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη τη ε, πραγματική οικονομία, πραγματική οικονομία σημαίνει εσωτερική αγορά, μικρομεσαίε επιχειρήσει και βιομηχανική πολιτική. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει χρειάζονται καινοτομία. Πρέπει να ε, γίνουν καινοτόμε για να ανταγωνιστικές και στην εσωτερική αγορά, αλλά και στις ε, εξοκοινωτικές αγορές. Και χρειάζονται, όπως είπε και ο κύριος Μπουσόη, να έχουν πρόσβαση στην ε, πίστη, σε δάνεια, στις κεφαλαγορές. Γιατί η καινοτομία για μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να γίνει με τα δικά της μέσα, αλλά για μια μικρομεσαία επιχείρηση, αν θέλει να αλλάξει, να αναπτύξει καινοτομία, πρέπει να υποστηριχθεί από μέσα εξωτερικά. Προσπαθούμε να τροποποιήσουμε με την, ε, μαζί με την Επίτροπο Γεώργιν Κουίν τα, όλο το πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ περίπλοκη η όλη διαδικασία. Όταν ήμουν ε, Επίτροπος Μεταφορών, ε, προώθησα το Μάρκο Πόλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το κάναμε επίσης και κάναμε μια προσπάθεια ως Επιτροπή με τον κανονισμό REACH. Ε, αφορούσε αυτό την ε, καταχώρηση. Μειώσαμε κατά 90% τους, ε, τα τέλη καταχώρησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια του REACH. Την περασμένη εβδομάδα συνέβη κάτι που γνωρίζετε δημιουργήθηκε αυτό το φόρουμ, ε, συγκαλέστηκε μάλλον αυτό το φόρουμ για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πίστοση. Και στην τελευταία συνεδρίαση που συμμετείχα, και αυτό είναι σημαντικό ε, μήνυμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για πρώτη φορά συμμετείχε ένας Βρετανός, ένα Βρετανικό διευθυντικό στέλεχος, ε, ο οποίος μας μίλησε για το θέμα της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην ε, πίστοση. Μας είπε, υπάρχουν τα λεφτά. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σχέδιο από τον κόσμο του, των χρηματαγορών για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. αυτή η δήλωση είναι σημαντική. Γιατί όταν ο κόσμος του χρήματος, όταν ας πούμε το χρηματιστήριο του Λονδίνου αποφασίσει να συνταχθεί υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημαίνει ότι το κλίμα για την πραγματική οικονομία αλλάζει. Εγώ δεν είμαι εναντίον των τραπεζών ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ε, λέω απλώς ότι τράπεζες και κεφαλαιαγορές, χρηματαγορές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία. Έχουμε τα κονδύλια του 7ου και 8ου προγράμματος πλαίσιο και έχουμε τα κονδύλια από ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν υπέρ της πραγματικής οικονομίας. Στα πλαίσια της δουλειάς που θα κάνουμε για την τυποποίηση, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε σύντομα συγκεκριμένες απαντήσεις Εδώ απαντάω και στον κύριο Κορέντε κάπως και στον κύριο Σβάπ για την τυποποίηση των οχημάτων των ηλεκτρικών, την τυποποίηση μάλλον των ηλεκτρικών ε, οχημάτων. Πέρυσι έδωσα εντολή στο ΣΕΝΕΛΕΚ για να προωθήσει αυτό το θέμα πριν το τέλος του 2011. Για τα ηλεκτρικά οχήματα έχουμε κανόνες ό,τι αφορά την ηλεκτρική ασφάλεια και η Κομισιόν πρότεινε να είναι δεσμευτικοί αυτοί οι κανόνες για την τυποποίηση των ε, ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης, τροποποιήθηκαν οι κανόνες UNESE για να καλύψουμε και συγκεκριμένους κινδύνους που αφορούν ειδικά τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι κανόνες για τα, την ηλεκτρική ασφάλεια και την ασφάλεια σε περίπτωση σύγκρουσης θα ληφθούν υπόψη για την ε, τυποποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων από την 1η Νοεμβρίου του 2012 για τα νέα οχήματα και από την 1η Νοεμβρίου του 2014 για τα οχήματα πάλι νέα, λέει ο Επίτροπος. Σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια, εγώ ε, υποστηρίζω το σήμα CE. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν και τη στιγμή της εισαγωγής των προϊόντων και μετά όμως, δηλαδή όταν τα προϊόντα μπουν στην εσωτερική αγορά. Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μια υπηρεσία τελωνιακή δική της, δεν έχει αστυνομία δική της που μπορεί να ελέγχει την αγορά. Επομένως θα πρέπει να εμπιστευτούμε άλλους, να υπάρξει συντονισμός, να υπάρχει συνεργασία και αυτή η άλλη φυσικά είναι τα κράτη-μέλη. Επομένως πιέζουμε τα κράτη-μέλη, στηρίζουμε τα κράτη-μέλη ε, δουλεύουμε και για το θέμα των ε, λιμένων που διαχειρίζονται τρίτες χώρες. Εκεί θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι ακριβώ κανόνες. Για το βασικό θέμα του ελέγχου, εδώ ε, συνεργαζόμαστε με τελωνία διαφόρων χωρών, γιατί από εκεί μπαίνουν πολλά ε, ξένα προϊόντα. Παραδείγματο χάρη το λιμάνι του Ρότερνταμ, που είναι το πιο σημαντικό λιμάνι στην Ευρώπη. Επομένω, είναι σημαντικό να γίνονται έλεγχοι εκεί. Εγώ σκοπεύω να πάω τον Ιούλιο και επιτόπου, για να δω πώς ετοιμάζονται οι αρχές για να τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία για τα παιχνίδια, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουλίου. Θα επιμείνω λοιπόν τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν, ούτω ώστε να εγκρίνουν τους ε, κανόνες για τη μεταφορά αυτής της οδηγίας για το θέμα του Εύρυκα. Ε, εγώ πάντα είμαι υπέρ όλων των πρωτοβουλειών, υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την αναθεώρηση του Small Business Act, έχουμε τον ε, κύριο Ντανιέλ Καγέχα, υποδιευθυντή, συγγνώμη, γενικό διευθυντή στη Γενική μου Διεύθυνση, ε, κάνει ο κύριος αυτός επισκέψει στις διάφορες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση για να δούμε πώς υποδέχονται το Small Business Act. Πήγαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, στην Ιταλία, θα πάμε στη Βουλγαρία ω τον Ούπο. α, πήγαμε και στη Γαλλία. Κάθε φορά που, πάω σε μια χώρα, που πάει εκείνο σε μια χώρα για να παρουσιάσει το Small Business Act, τον συνοδεύω. Γιατί τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να διορίσουν, όπως ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα πρέσβη για την εφαρμογή του Small Business Act στη συγκεκριμένη ε, χώρα, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Ευρωπαίο πρέσβη για αυτό το θέμα. Κάθε χρόνο θα συνέρχονται όλοι οι πρέσβεις όλων των διαφορετικών ε, κρατών μελών με τον Ευρωπαίο πρέσβη, με τον πρέσβη δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα που θα μιλήσει αποκλειστικά για το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο τελευταίο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα, όλοι κατά τη διάρκεια του γεύματο είπαν ότι είναι υπέρ αυτή τη ιδέα. Ορισμένε χώρε έχουν ήδη διορίσει αυτόν τον πρέσβη. Η Ιταλία έχει διορίσει έναν διευθυντή του Υπουργείου Οικονομική Ανάπτυξη. Η Γαλλία θα τον διορίσει τώρα αυτόν τον πρέσβη. Η Μάλτα έχει προβλέψει το διορισμό του στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Small Business Act. Έτσι μου είπε ο υπουργό στο τελευταίο Συμβούλιο. Η Ισπανία την περασμένη εβδομάδα διόρισε επευκαιρία της παρουσίας του Small Business Act στη Μαδρίτη με τον Υπουργό τον κύριο Σεμπαστιάν. Ε, διόρισε μία πρέσβυρα μάλιστα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια κυρία. Αρχίζει λοιπόν να υλοποιείται όλη αυτή η ιστορία και σε επίπεδο κρατών μελών. Συζητήσαμε με τον Υπουργό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου σε μία συνεδρίαση όπου ήταν και ο πρόεδρος ο κ. Χάρμπουρ, ούτως ώστε όλες οι χώρες να κάνουν ε, πράγματα υπέρ της επιχειρηματικότητας. Με μεγάλη χαρά σημείωσα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει μία προσπάθεια υπέρ της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, υποστηρίζοντας έντονα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως τις καινοτόμες. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί από έναν Ευρωπαίο Επίτροπο, με μεγάλη χαρά μάλιστα, γιατί όταν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρωταγωνιστή για την ανάπτυξη τη ε, πραγματική οικονομία, αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα και πρέπει να τονιστεί. Well, we very much χαιρετίζουμε ότι ταξιδεύεται και σε ευρύ πλαίσιο και την οδηγία για τα παιχνίδια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία τώρα. Διότι τα παιχνίδια για τα επόμενα Χριστούγεννα θα, ξεκινούν, θα ξεκινήσουν να παράγονται σύντομα. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα πιέζει πολύ ο χρόνο. Θα ζητήσω από τους απομείναντες αγορητές 6-7 στον κατάλογο. Πολύ σύντομη να είσαστε στη διατύπωση των ερωτήσεων σας. Πιέζει ο χρόνος, λυπάμαι. Χώσιτς, Ρούλε, Στάιλερ, Άμπατ, Μικρύπ, η κυρία Ράπτη και ο κύριος Μπουσουτήρ. Λοιπόν, ένα λεπτό καθένας, έτσι, συνολικά. Θα έχει πολύ λίγο χρόνο στη συνέχεια να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ας το προσπαθήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ας δοκιμάσουμε. Κόζονικ πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο, ε, λέγει ο κύριος ε, Κόζοτσικ. Κύριε ε, Επίτροπε, χαίρομαι γιατί τακτικά παρακολουθείτε συνεδρία τη Επιτροπή μα και θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στη συνέχεια για τη δουλειά που αναπτύσσεται σε σχέση με την νομοθεσία, νομοθετικές προτάσεις για την τυποποίηση και τις ενιαίες προδιαγραφές και ελπίζω ότι πολύ προσεκτικά θα ακολουθηθεί και η δική μας η γραμμή από πλευρά σας συνολικά ότι δεν θα υπάρξει κάποια ανατροπή επανάσταση εδώ, αλλά θα είμαστε συνεπείς. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συνεργασία με τους υπεύθυνου του γραφείου σας, της υπηρεσίας σας. Μια συγκεκριμένη ερώτηση έχω, αφορά ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει. Είναι το σύστημα Γαλιλαίος αυτό το θέμα συγκεκριμένες πληροφορίες ε, για την μεταφορά της διαχείρισης ε, και ε, ελέγχου του συστήματος στην Πράγα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με την Τσεχία και πότε η μεταφορά αυτή του Γαλιλαίου θα ολοκληρωθεί σε σχέση με την Τσεχία. Ευχαριστώ will allow Ειδική ερώτηση. Δεν βρίσκεται στις, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, αλλά παρόλα αυτά, αυτή είναι η ερώτησή σα, η κυρία Ρούλε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα προσπαθήσω να αποφύγω επαναλήψεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έγιναν ήδη. Καταρχήν ευχαριστώ για την καλή συνεργασία για τα οικοδομικά υλικά και προϊόντα. Έχουμε ένα καλό κανονισμό που έχει εγκριθεί. Τι θα γίνει με τις κατεντολήν πράξεις στη συνέχεια, την εντεταλμένη αυτή και με τις, ε, για τις ε, οερονόμ, τις ευρωπαϊκές ε, διατάξεις. Καθώς επίσης και σε σχέση με τις συμβάσεις το πρόβλημα είναι της καινοτόμας διαδικασίας για τις ηλεκτρονικές προμήθειες. Τι μπορεί να γίνει ώστε να ενημερώνονται τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτό και μία άλλη ε, πτυχή, η εποπτεία της αγοράς. Ε, σε σχέση με την επαναδιατύπωση της ασφάλειας των προϊόντων και ενιαίοι ε, έλεγχοι και συστήματα ελέγχων σύμφωνα με την εμπειρία σε σχέση με τα κράτη-μέλη αντί να αυξηθούν μειώνονται περισσότερο. Δεν θα μπορούσαν εδώ ελάχιστες προδιαγραφές να θεσπιστούν για την εποπτεία της αγοράς και η τελευταία ερώτηση και που αφορά και τα θέματα των παιχνιδιών. Την ερώτηση του κ. Σουβάπ δεν την απαντήσατε. Έχουμε το πρόβλημα στα κράτη-μέλη στην υλοποίηση, στην εφαρμογή όταν οι οριακές τιμές ε, πρέπει να μειωθούν, να, χαμηλώσουν και μετά να αυξηθούν σε μια επόμενη φάση. Δεν μπορούμε πιο γρήγορα να πορευτούμε με τη διαδικασία επιτροπολογίας. Ευχαριστώ. Τέσσερις ερωτήσεις σε 1,5 λεπτό είναι πραγματική επίδοση. Η κυρία Στάιλερ, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ Επίτροπε, για την εποπτεία της αγορά. Θα ήθελα να κάνω την παρατήρηση για το γεγονό ότι οι προπολογισμοί των κρατών μελών έχουν περιοριστεί και προφανώς σε σχέση με τι οργανώσεις που αναλαμβάνουν την εποπτεία στα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η δουλειά θα μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των κρατών μελών συμφωνώ μαζί σας σε σχέση με την καινοτομία στις ε, ε, αγορές και προμήθειες. Γιατί δεν υλοποιείται αυτή η οδηγία όμως ε, για τα παιχνίδια από βράσκα των μελών. Και για αυτό που είπε η κυρία Ρούλε για τη σημασία του οικοδομικού τομέα. Και έχουμε σε σχέση με αυτό συζητήσει και την δυνατότητα μέσα σε μια ετήσια συζήτηση να δούμε τι μπορεί να γίνει. Διαρωτώ με, Έχετε θετική προσέγγιση για αυτή την πρωτοβουλία, για να προσεγγίσουμε αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ. Αμπάντ, παρακαλώ, επόμενος αγορητής. Oui, merci, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε και συγχαρητήρια. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα, Small Business Act και η σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Δύο πράγματα. Θα ψηφιστεί νομοθεσία για εργολάβους, εργολήπτες δηλαδή, και αυτούς που δίνουν τις εντολές. Θα υπάρξουν ρυθμίσεις στον τομέα αυτό. Επίσης, ως πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για την ε, Νεολαία, θα κάνετε κάτι για τον έρασμο που μας ε, απασχολεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Η ερώτησή μου είναι απλή. Και έρχομαι στην ουσία. Από κοινού με τον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ ανακοινώσατε την ανάληψη πρωτοβουλίας για επενδύσεις εκτός Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο τρόπο θα γίνει η αξιολόγηση των επιπτώσεων ορισμένων επενδύσεων που προέρχονται από έξω από την Ευρώπη στην Ευρώπη σε ορισμένους τομείς της οικονομίας μας και της βιομηχανίας. Η κυρία Ράπτη, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα περισσότερα ζητήματα καλύφθηκαν. Α, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την δουλειά που σχεδιάζει σε σχέση με τα παιχνίδια. Και το επισημαίνω αυτό γιατί ήμουν από αυτούς που το Δεκέμβριο στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια είχα βάλει τις φωνές. Ε, έτσι λοιπόν ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνει. Θα είμαστε βέβαια πάντα εκεί το Δεκέμβριο για να δούμε τα αποτελέσματα, αλλά ως ένδειξη καλής θέλησης δίνω το υπόλοιπο του χρόνου μου για να απαντήσει. Κύριος Μπουσουτήλ, τελευταίος παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο Ταγιάννη για όσα είπε για μια νέα νομοθετική πρόταση για την καταχώρηση των αυτοκινήτων και τα τέλη των φόρων σχετικά με την τάξη νόμιση. Θα ήθελα να ρωτήσω τι έγινε σε σχέση με την νομοθετική πρόταση επί του ιδίου θέματος που στόχευε σε έναν εναρμονισμό ή σε κάποιο είδος εναρμονισμού σε αυτό το τομέα που είχαμε υπερψηφίσει πριν από 3-4 χρόνια ως πρόταση. Αυτή η σε καποιο ειδος εναρμονισμου σε αυτο το τομεα που ειχαμε υπερψηφισει πριν απο τρια η 4 χρονια ως προταση αυτη η προταση για αυτή την πρόταση δεν ξανακούσαμε τίποτα πια μετά. Δεν ξέρουμε αν ε, λίμνασε, αποτελματώθηκε στο Συμβούλιο ή τι συμβαίνει με την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι περιορισμένο ο χρόνο, έχουμε 5-7 λεπτά. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να προσπαθήσετε να απαντήσετε και λεπτομερεί απαντήσει να δοθούν στη συνέχεια. Για την οδηγία για τα παιχνίδια, ε, θέλω να προχωρήσουμε με βάση το χρονοδιάγραμμα. Και κυρίως για τις επικίνδυνες ουσίες, για το κάδμιο και Μόλιβδο, θα προχωρήσουμε. Για τα κατασκευαστικά έργα. Κυρία Ρούλε, σας είχα υποσχεθεί ένα οδικό χάρτη για την εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα, για τον κατασκευαστικό τομέα. Θα την έχετε ως ονούπο αυτή την πρόταση. Σε ό,τι αφορά τώρα την εποπτεία της αγοράς, Πρέπει να επαναλάβω αυτό που σας είπα. Μπορούμε να έχουμε ωραιότατους κανόνες, αλλά τα κάτι μελη πρέπει να, του, να τους εφαρμόζουν. Δεν έχουμε τα μέσα για να ελέγξουμε. Εγώ μπορώ να δώσω το παράδειγμα. Να πάω στο Ρότερνταμ, μας πούμε, και να πω, να, ορίστε, εδώ, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Όταν αποφασίσουμε να αποκτήσουμε το δικό μας, τα δικά μας τελωνία και τη δική μας αστυνομία θα κάνουμε και αυτοπροσώπους ελέγχους. Αλλά κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε. Ε, για το έρασμος, για τους νέους επιχειρηματίες θα προχωρήσουμε. Είναι ανοιχτή συζήτηση και για τον προπολογισμό της επόμενης χρονιάς, αλλά και για τις οικονομικές ε, προοπτικές. Και η υποστήριξη του Κοινοβουλίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι θεμελιώδης, είναι εκ των όνου για να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε αυτά τα παράθυρα για όλους τους τομείς, ούτως ώστε πέρα από την οριζόντια δράση να έχουμε στα πλαίσια κάθε γενικής διεύθυνσης μία σημαντική δράση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα, για το Γαλιλαίο. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γαλιλαίος δεν πρέπει να είναι μόνο ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την Ιταλία, η Γερμανία και τη Γαλλία, τις χώρες που έχουν σχετική βιομηχανία αεροναυπηγικής θα πρέπει να αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Είμαι για την σημασία αυτή της ε, υπηρεσίας ε, η οποία θα εδρεύει στην Πράγα. Είναι σημαντικό. Την περασμένη εβδομάδα υπέγραψα στη Μαδρίτη μια συμφωνία με την Ισπανική κυβέρνηση για να δημιουργήσουμε στη Μαδρίτη την τρίτη έδρα, μια ε, στην Ιταλία, μια στη Γερμανία και μια στην Ισπανία για τις υπηρεσίες, η τρίτη δηλαδή. Ε, στο τορεχόν. Εκεί θα εδρεύει αυτή η υπηρεσία. Για το ερώτημα της κυρίας Γκριπ, για τις επενδύσεις από το εξωτερικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συζήτησα με τον Επίτροπο Μπαρνιέ για ένα πρόβλημα που υπάρχει Φυσικά απόκειται στον πρόεδρο να αποφασίσει αν είναι σκόπιμο να το φάλει στη μέση διάταξη της Κομισιόν και να πάρουμε μια απόφαση ως Κομισιόν. Εγώ είμαι πολιτικός και αντιμετωπίζω πολιτικά προβλήματα. Πάντως να είναι ξεκάθαρο το εξή. Εμείς δεν έχουμε καμία προστατευτική θέση. Είμαστε σαφώς υπέρ της ανάπτυξη των επενδύσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και όταν οι επενδύσεις αυτές προέρχονται από φορείς, από άτομα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ευπρόσδεκτες οι επενδύσεις στην Ευρώπη. Το μόνο πρόβλημα που θέσαμε αφορά την προστασία του know-how, savoir-faire, τεχνογνωσία, το λέω σε όλες τις γλώσσες, που είναι το εργαλείο για να εξασφαλίσει ε, ανταγωνισμό ε, ποιότητας η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κανένα προστατευτισμό λοιπόν, απλώς προστασία. Όχι προστατευτισμό. Γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ξένα συμφέροντα ε, αυτών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το δικό μας know-how τη δική μας πραγματογνωμοσύνη για να την ε, εξάγουν από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι λιγότερο ακριβό να αγοράσεις όλη τη βιομηχανία, μια βιομηχανία, έτσι, με το know-how της και μετά την κλείσει. παρά να ξεκινήσεις έρευνα και έρευνα και καινοτομία σε μια άλλη χώρα από το μηδέν. Στην Ιταλία, τη χώρα μας, υπάρχει μια έκθεση της κυβέρνησης που υποβλήθηκε στην Ιταλική Βουλή των Μυστικών Υπηρεσιών, που λέει ότι υπάρχει μια δράση από βιομηχανικούς τομείς ξένους στο εξωτερικό για να αγοράσουν και να εξάγουν από την Ευρώπη το know-how της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ο Επίτροπος Βιομηχανίας εγώ δηλαδή που είμαι και Ευρωπαίος πολιτικός, πρέπει να θέσει αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορώ εγώ να πάρω την απόφαση. Αλλά στην Κίνα και στην, στη ΣΥΠΑ υπάρχουν συστήματα ελέγχου για του στρατηγικούς τομεί. Έτσι. Ε, αυτό που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κανόνες. Εγώ και ο Επίτροπος Μπαρνιέ θέσαμε αυτό το πρόβλημα υπόψη έξι υπουργών. Ε, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Πολωνία. Υπάρχει και ένα άρθρο στην Μόντα ε, για αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να πάρω σχετική απόφαση, αλλά νομίζω ότι είναι καθήκον μου και για να υπερασπίσω την, υπερασπίσω την ε, εσωτερική αγορά ως Επίτροπος Βιομηχανίας να γνωστοποιήσω αυτό το πρόβλημα στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα θεμελιώδου σημασίας για την ε, οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μια επιλογή προστατευτισμού. Το διαψεύδω όποιο είπε κάτι τέτοιο, γιατί είμαι πραγματικά υπέρ των ξένων επενδύσεων. Απλώ δεν θέλω να αγοράσουν το know-how μα, ε, ειδικά κάποιων στρατηγικών ε, βιομηχανικών τομέων, και να το εξάγουν. Μάλιστα, τώρα, σε ό,τι αφορά την καταχώρηση των αυτοκινήτων. Με βάση τα δεδομένα στο παρελθόν, τα δεδομένα του παρελθόντος Πρέπει να προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση καταχώρηση. Σε ό,τι αφορά το, αίτημα, το ερώτημα του κ. Μπουσουτή, δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποια είναι η κατάληξη αυτής της πρότασης. Ε, δώστε μου λίγο χρόνο και σε 24 ώρες θα σας απαντήσω πιο συγκεκριμένα στο ερώτημα. Να, για να δω τι κατάληξη έχει αυτή η πρόταση στην οποία αναφερθήκατε. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις απαντήσεις. Πάντως είμαι στη διάθεσή σας και για περαιτέρω ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Ξέρετε ότι είμαι πάντα έτοιμος να ε, συναντήσω βουλευτές. Και στο Στρασβούργο έχουμε και μία φορά κάθε Στρασβούργο, εν πάση περιπτώσει, είμαι εκεί για να έρθω σε επαφή με βουλευτέ κτλ. Μπορώ να σας δώσω και τεχνικές διευκρινήσεις ώστε να μπορέσετε να δουλέψετε καλύτερα. Ευχαριστώ. Uh, Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Αντώνιο, κύριε διπρόεδρε, που αντιμετωπίσατε θαραλέα όλες αυτές τις ερωτήσεις. Είναι διεξοδικό το πρόγραμμα εργασιών σας. Ίσως μπορεί η ομάδα των συνεργατών σας να μας υποβάλει μια σύνοψη των αναμενωμένων, γιατί ε, θα μπορούμε να τα αποκριθούμε καλύτερα έτσι. Βεβαίω θα παραμείνουμε σε διάλογο μαζί σας και τον επόμενο χρόνο αλλά και ε, στο υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής θητείας. Έχετε στο χαρατοφυλάκιο, σας πολλά θέματα που είναι σημαντικά για την Επιτροπή μας. Για παράδειγμα ασφάλεια προϊόντων, λειτουργία της ενίας αγοράς, η αναμενόμενη νέα τεχνολογία αυτοκινήτων. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε, ευχαριστώ και, τους, και τις και τους Γερμηνείς που παρέμειναν μαζί μας λίγο περισσότερο. Θα συνεδριάσουμε ξανά δημοσίως το απόγευμα στις 4.30. Έχουμε ακρόαση για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα, για να το πω επισήμως, δηλαδή μοτοσυκλέτες και άλλα σχετικά. Θα κάνουμε ακρόαση με συμμετοχή του εισηγητού κ. Βαντεκάμπ στις 4.30 λοιπόν, οι δε συντονιστές των κοινοβουλευτικών ομάδων θα συναντηθούν μαζί μου στις 3. Διακόπτω τη συνεδρίαση.